Alle, Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σα. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει όλοι να αισθανόμαστε πολύ περήφανοι που ήρθαμε εδώ τόσο πρωί. Είστε, είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι, δεν έχουμε θέματα ημερήσιας διάταξης, δεν έχω ανακοινώσει Προέδρου και άρα μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στο πρώτο θέμα ε, και θέλω να καλωσορίσω τον Πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου, τον κύριο Τουκάνοβιτς. Είμαστε πολύ ευτυχείς που βρίσκεστε εδώ. Για πρώτη φορά έχετε έρθει στην Επιτροπή μας. Έχετε αναλάβει διάφορες ευθύνες τα τελευταία 25 χρόνια στη χώρα σας και τώρα έχετε ενώπιόν σας προεκλογική εκστρατεία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 Drittstaaten. Wir Λοιπόν, είστε μια σημαντική τρίτη χώρα. Σας ευχόμαστε θάρρος, δύναμη, κουράγιο για να αντιμετωπίσετε τα θέματα και να, ε, περάσετε, να περασπιστείτε τα συμφέροντα της χώρας σας. Θα σας δώσω το λόγο για να μας μείνει επαρκής χρόνος και για συζήτηση. Poštovani gospodine Κύριε Μπροκ, μέλη του Κοινοβουλίου, μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά τιμή και χαρά για μένα που σας συναντώ εκ μέρους της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου. Η σημερινή μας συνάντηση επιβεβαιώνει την αφοσίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία της διεύρυνσης και μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα του Μαυροβουνίου εν ώψη των διαπραγματεύσεων των ε, ε, ένταξης και τις επόμενες φάσεις. Ε, φέτος είναι μια σημαντική χρονιά και γιατί έχουμε την επέτειο της ανεξαρτησίας μας, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε προχωρήσει καλά, έχουμε υπόψη μας την σύνταξη του Κοινοβουλίου, τη σύνταξη της έκθεσης για το Μαυροβούνιο το 2016 που θα δημοσιευτεί μετά τις εκλογές. Πιστεύουμε ότι οι εκλογές που θα γίνουν φέτος θα προωθήσουν τον διάλογο και την συμφωνία όπως ε, διατυπώνονται στην ε, συμφωνία κυβέρνηση με το μεγαλύτερο μέρος αντιπολίτευσης για τις δίκαιες εκλογές. Πιστεύουμε ότι από εδώ και πέρα θα χαρακτηριστεί η πολιτική μας ζωή ζωή ε, από μια νέα φάση όπου θα υπάρχει συνεπής κοινοβουλευτική ε, πλειοψηφία και θα οδηγήσει σε, δημοκρατικές, ε, σε ανάπτυξη δημοκρατία. Η SAPC και το ψήφισμα για το Μαυροβούνιο πιστεύουμε ότι θα αναφερθούν στα θετικά αποτελέσματα της συμφωνίας ε, αφορούν την κυβέρνηση για την εκλογική εμπιστοσύνη. Όπως θα γνωρίζετε, κάλεσα την, κάλεσα την αντιπολίτευση να συνεργαστεί με την κυβέρνηση και τους προσέφερα βασικά υπουργεία όπου θεωρούν ότι γίνεται κατάχρηση των ε, κρατικών πόρων υπέρ των εκλογών, δηλαδή Υπουργείο Οικονομικών, Εσωτερικών, Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Από φέτος έχουμε επικεφαλής των Υπουργείων αυτών από την αντιπολίτευση. Έχουν επίσης δεχτεί να αναλάβουν τη θέση, μια θέση αναπληρωτή ε, πρωθυπουργού στην κυβέρνηση. Επίσης σε όλα τα επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοσίων επιχειρήσεων έχουν εκπροσώπους. Η ιδέα ήταν να επιδιώξουν ψάξουμε λύσεις ε, για τα προβλήματα που βαρύνουν την πολιτική μας ζωή μέσω διαλόγου με τα θεσμικά όργανα. Έχουμε ξεπεράσει την ε, ε, δυσπιστία που είχαν δείξει οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης για τα εκλογικά αποτελέσματα και αυτό συνέβη μετά από την εποχή ήδη του ε, δημοψηφίσματος και την ανεξαρτησία. Σας διαβεβαιώ ότι οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι σημαντικές και αντικειμενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη χώρα μας, την πορεία της ένταξης. Είμαστε ιδιαίτερως ευγνώμονες ε, για την, το ενδιαφέρον και την υποστήριξή σας, όπως επίσης την αναγνώριση της ποιότητας της δουλειάς μας στον δρόμο μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην δύσκολη αυτή περίοδο που αντιμετωπίζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να πούμε ότι η ενοποίηση στην πολυφωνία είναι ε, εξίσου σημαντική και τώρα. Αυτή η ενοποίηση στα πλαίσια της Ευρώπης αποτελεί σημαντικό κίνητρο να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις και να θεσπίσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο επιδιώκει την επίτευξη των ευρωπαϊκών αρχών και θεωρούμε ε, την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικό ε, στόχο της εξωτερικής μας πολιτικής. Υπάρχει ε, υποστήριξη κοινή γνώμης προς αυτή την κατεύθυνση. Η ένταξη είναι σημαντικός παράγων της οικονομικής και, σταθε... και δημοκρατικής σταθερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια. Η περαιτέρω πρόοδος των σχέσεων του Μαυροβουνίου με τους γείτονες σε σχέση με την ενωμητάξη και την ενίσχυση των υποδομών τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις ξένες επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελεί το βασικό κίνητρο όλων μας. κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις της ένταξης για να εξασφαλίσουμε μια γενικότερη οικονομική αλλαγή και να εκπληρωθούν οι όροι της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας ένα σημαντικό στοιχείο είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ που επίκειται υπάρχει και που θα επηρεάσει θετικά την ευρύτερη περιοχή. Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα της πορείας ένταξης εγγυώνται τις μελλοντικές επιτυχίες. Το άνοιγμα των 24 κεφαλαίων της διαπραγμάτευσης η αλλαγή και η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και τα κίνητρα για την ε, ανάπτυξη υποδομών Πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές με βιώσιμο τρόπο. Αυτό θα νομιμοποιήσει και τις περαιτέρω φάσεις της διαδικασίας για να είμαστε εντελώς έτοιμοι για ένταξη. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε νέα κεφάλαια πριν το τέλος του χρόνου, έχοντας υπόψη μας το ποσοστό της εκπλήρωσης των συγκριτικών δικτών και της θέσεις που έχουν διατυπωθεί για 29 κεφάλαια. Η, η ένταση, η εντατικοποίηση της δουλειάς μας για τις κοινέ θέσεις είναι κομμάτι των προσδιοκιών μας στα πλαίσια της ε, ε, διαπραγμάτευσης πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια της Σλοβακικής Προεδρίας και πολλών άλλων θα μπορέσουν να ανοίξουν και άλλα σημαντικά κεφάλαια. Ελπίζουμε στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών εταίρων ώστε να αρχίσουν να κλείνουν κάποια από τα πρώτα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων ως ένα ε, σύμβολο στήριξης της διαδικασίας της ε, διαπραγμάτευσης και του θετικού της αποτελέσματος. Αυτό είναι σημαντικό για την προώθηση των συνεπών ε, ε, κατευθυντηρίων γραμμών με, που έχουν αποφασιστεί με τους Ευρωπαίους συνομιλητές μας. Όλα αυτά έχουν σημασία και για τις ε, άλλες χώρες περιοχής μας. Αν είμαστε αφοσιωμένοι στην ε, θέσπιση των, του Ευρωπαϊκού συ, Συστήματος Αξιών, αυτό γίνεται σεβαστό από την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητες. Δίνουμε έμφαση στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τα κεφάλαια 23 και 24 που αφορούν τη νέα προσέγγιση και την εκπλήρωση των 83 ενδιάμεσων συγκριτικών δικτών. Η έκθεση του Απριλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι το Μαυροβούνιο βρίσκεται σε καλό δρόμο για την εκπλήρωση των συγκριτικών δικτών με περαιτέρω συστάσεις για δράση. Επίσης σημειώθηκε πρόοδος και κατά την ε, ε, ε, ε, εξαμηνία έκθεση της κυβέρνησης τα κεφάλαια 23 και 24. Η νομοθεσία έχει προχωρήσει, έχουμε περάσει πάνω από 60 νόμους από το Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι φέτος, του, μέχρι φέτος τον, το καλοκαίρι. Ήδη οι αλλαγές ε, σημειώνονται και βελτιώνουν ε, τις επιδόσεις μας. Η αποτελεσματικότητα και η αφοσίωση ε, φαίνονται και από το γεγονός ότι έχουμε ξεκινήσει έρευνες, έχουν γίνει δικαστικές αποφάσεις και έχει γίνει κατάσχεση περιουσιών αξίας άνω των 23 εκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση έχει αφοσιωθεί στην εκπλήρωση όλων των ενδιάμεσων δικτών των κεφαλαίων 23 και 24 και μας είναι σημαντικό γιατί το θέμα της ένομης τάξης είναι σημαντικός παράγοντας ασφάλειας για τους πολίτες μας. Συνεπώς λοιπόν ειδικά σε αυτόν τον τομέα θα δαπανίσουμε την περισσότερη ενέργεια την οποία έχουμε. θα υπογραμμίσουμε όχι τόσο την ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων όσο την ποιότητα των μεταρρυθμίσεων. Έχουμε ένα περίπλοκο περιβάλλον στην χώρα και στην περιοχή και γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία των πολιτικών εξελίξεων. Να συνειδητοποιούμε επίσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα, το Brexit, τη μετανάστευση, Όλα αυτά ε, ενθαρρύνουν κάποιες δυνάμεις ε, οι οποίες λειτουργούν αντιευρωπαϊκά. Και γι' αυτό ακριβώς ε, νομίζω ότι θα πρέπει να εμείνουμε και εμείς σαν χώρα στο υπάρχον ευρωπαϊκό πλαίσιο, στα πλαίσια και της πλειοψηφούσας άποψης στην Ευρώπη. Υπογραμμίζουμε λοιπόν για μια ακόμη φορά την μεγάλη ανάγκη συνεχούς ευρωπαϊκής υποστήριξης στην περιοχή μας. Η απόκτηση περαιτέρω ευρωπαϊκών χαρακτηριστικών στα Δυτικά Βαλκάνια είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν είναι θέμα συζητήσεων ή διαπραγματεύσεων, αλλά συνέχισης της προσπάθειας σταθεροποίησης της περιοχής, υιοθέτηση και αφομοίωσης των ευρωπαϊκών επιπέδων προστασίας του πολίτη και όλα αυτά θα παίξουν ρόλο όχι μόνο για μας αλλά και για την ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης. Ε. Έχουμε λοιπόν μια νέα εικόνα για τα Δυτικά Βαλκάνια στην περιοχή μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης να προχωρήσουμε σε περαιτέρω περιφερειακή συνεργασία, στη βελτίωση των υποδομών, έτσι ώστε να συνδεθούμε και με τους λεγόμενους ευρωπαϊκούς διαδρόμους. Έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και για την ενίσχυση του κράτους του δικαίου και της δημοκρατίας. Στον οικονομικό τομέα εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης, την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τα 10 χρόνια μετά την ανεξαρτησία είχαμε μέσο όρο οικονομικής ανάπτυξης τον χρόνο 3,2%. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2018 να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της χώρας μου και να προσελκύσουμε περαιτέρω ξένες επενδύσεις εκμεταλλευόμενοι το δυναμικό το οποίο παρέχει η χώρα μου και στα πλαίσια των συνεργασιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον τομέα της ενέργειας Νομίζω ότι όλες οι προσπάθειες αυτές θα μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμεθα. Θα διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και στον τομέα της φορολογίας. Όλα αυτά είναι εγγύηση για το μέλλον. Νομίζω ότι θα καταστούμε ακόμα πιο αξιόπιστο περιβάλλον οικονομικό. Εμείς προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα με υπευθυνότητα. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στην περιοχή μας, να καταστήσουμε την περιοχή μας μια ασφαλέστατη περιοχή, η οποία να είναι αφιερωμένη θα έλεγα, ή αφοσιωμένη συγγνώμη καλύτερα, στις προσπάθειες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό θα κάνει και τους πολίτες μας να πιστέψουν στην Ευρώπη ακόμα περισσότερο οι δραστηριότητές σας, οι δραστηριότητες του εισηγητή σας, του κύριου Τάνοκ, οι δραστηριότητες της κυρίας Ντόντς, όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά για, το Μαυροβούνιο και οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας βοηθούν και μας καθοδηγούν στην πορεία για, την, για τον ευρωπαϊκό στόχο. Ε, φυσικά και εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τον διάλογο μαζί σας ώσπου να πετύχουμε να γίνουμε πλήρες μέλος. Νομίζω ότι το Μαυροβούνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρότυπο ε, για την μελλοντική εξέλιξη της περιοχής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρωθυπουργέ για τα όσα μας εκθέσατε και από τη διερμηνία από τη γλώσσα σας τη γλώσσα του Μοντενέγκρο είναι στο 25 όχι στο 28 εν πάση περιπτώσει περνάμε στη συζήτηση τώρα ο συνάδελφος πρέπει να τον λόγο παρακαλώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Ευχαριστώ και τον κύριο Πρωθυπουργό. Τον ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ σήμερα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις με προσωπικότητες όπως εσείς για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Να συγχαρώ τη χώρα σας για την εξαιρετική πορεία στις διαπραγματεύσεις μέχρι σήμερα Λέγεται ότι είπατε μάλλον ότι θα ανοίξετε νέα κεφάλαια, οπότε θα συνεχίσετε την καλή αυτή πορεία. Να συγχαρώ το Μαυροβούνιο και για την υπογραφή του πρωτοκόλου συνεργασίας με τον ΝΑΤΟ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την περιοχή σας ιδιαίτερα να συνεργαστεί με τον ΝΑΤΟ. Και η χώρα σας συμμερίζεται τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξωτερική πολιτική και στον τομέα των κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας. Κάτι το οποίο δεν ισχύει πάντα. Τώρα για τη διαδικασία διεύρυνσης. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Η Ολλανδική Προεδρία δεν είπε τίποτα στο πρόγραμμά της για τη διεύρυνση. Η Σλοβακική Προεδρία επανήλθε στην διαδικασία αυτή. Χτες πάλι ο πρόεδρος Γιούγκερ, δεν βρήκε χρόνο να αναφερθεί έστω και μία φορά στα της διεύρυνσης. Ε, αυτή την κατάσταση εσείς πώς την βιώνετε, τι λέγετε στη χώρα σας, τι λέτε εσείς ο ίδιος για αυτές τις εναλλαγές θα έλεγα της χρήσης της έννοιας της διεύρυνσης στα θεσμικά όργανα. Κύριε <clears throat> uh, Πρόεδρε, καλώς ορίσατε θερμά Πρωθυπουργέ Τζουκάνοβιτς ε, και ως ε, ο εισηγητής για το Μαυροβούνιο. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια που αναφέρατε στο λόγο σας. Ε. Και έχω εδώ το αξίωμα για την αρμοδιότητα από πλευράς των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών που υποστηρίζουν πολύ τη διεύρυνση της Ένωσης με τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και πρέπει να πω, και αυτό είναι μια προσωπική δήλωση φυσικά, ότι είσαστε ένας ξεχωριστός πρωθυπουργός και περιφερειακός ηγέτης στα Δυτικά Βαλκάνια, ένας βετεράνος, παλέμαχος πραγματικά για τις μάχες ε, του Μαυροβουνίου μετά από 10 χρόνια ανεξαρτησίας ε, της χώρας σας και θέλω φυσικά να σας συγχαρώ και για την πρωτοβουλία σας που έχετε μια κυβέρνηση ολοκληρωμένη και από, πολλά, από, διάφορους, ε, διάφορες πολιτικές συνιστώσεις ε, και υπάρχει εμπιστοσύνη και χαίρομαι που συνεχίζεται αυτή η πορεία με σταθερότητα και με ικανοποιητικό τρόπο καταφέρνετε να διαχειριστείτε τις διαδικασίες ε, που βρισκόντουσαν υπό εξέλιξη και ήταν αποσταθεροποιητικές για το Μαυροβούνιο και σε σχέση με τον συνασπισμό στον οποίο είσαστε ένα τμήμα Επίσης για τη διαδικασία επικύρωσης που συνεχίζεται με θετικό τρόπο και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο και γνωρίζουμε ότι σίγουρα το Ηνωμένο Βασίλειο παρόλη την κατάσταση του Brexit της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση διμερώς υποστηρίζει το Μαυροβούνιο και τις προσπάθειές του. Κάπως ανησυχώ φυσικό ότι το μπλοκ της αντιπολίτευσης θέλει ένα δημοψήφισμα εφόλων αυτών υπήρξε εκστρατεία, τουλάχιστον για την πρόσφατη εκστρατεία στη χώρα μας όσον αφορά το Brexit, και έχω σημαντικές επιφυλάξεις πλέον για δημοψηφίσματα όσον αφορά τη ρύθμιση πολιτικών θεμάτων. Παρότι μπορεί να υπάρχουν ίσως κάποιες ενδείξεις ή τεκμήρια, γίνονται συναισθηματικά ιδιαίτερα φορτισμένα αυτά τα θέματα και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας τρόπος να, να διαχέονται, να διαβιβάζονται γεγονότα και τεκμήρια αντικειμενικά και σε σχέση με το ε, Μαυροβούνιο αν θα γίνει δημοψήφισμα για παράδειγμα για την προσχώρησή σας στο ΝΑΤΟ ή όχι καλωσορίζω τις πραγματιστικές παρατηρήσεις σας σε σχέση με το Κωσυφοπέδιο κάνατε πρόσφατα μια δήλωση για τον καθορισμό της μεθοριακής γραμμής της, ε, των συνόρων είναι ένας επιτυχής περιφερειακός παίκτη ε, το Μαυροβούνιο και πραγματικά μπορεί και προσπαθεί να μεσολαβήσει μεταξύ άλλων χωρών όταν αρχίζουν να υπάρχουν τριβές και οι σχέσεις επιδεινώνονται. Ελπίζω ότι το πρόβλημα του κοσυφοπεδίου και το θέμα των συνόρων θα μπορέσει σύντομα γοργά να ε, διευθετηθεί. Τώρα, σε σχέση με τις 16 ε, Οκτωβρίου θα γίνουν εκλογές, εκλογές που θα διεξαχθούν υπό ένα αναθεωρημένο, ευρύτερα αναθεωρημένο πλαίσιο, το καλωσορίζουμε αυτό, μεταξύ άλλων ε, αλλαγών και τις ε, αλλαγέ όσον αφορά τους συμβούλους και τους ε, κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους ένα ολόκληρο νέο σύστημα, νέες διαδικασίες για την καταχώρηση υποψηφίων και ιδιαίτερα και όσον αφορά υποψηφίους μειονοτικών λιστών, καταλόγων. Αυτά είναι νομίζω θετικά για τη χώρα σας. Και όπως και στις προηγούμενες εκθέσεις μου ανέφερα, μια και ήμουν μόνιμο εισηγητής για 7 χρόνια για αυτό το ζήτημα, είμαι νομίζω για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εισηγητής, μόνιμος εισηγητής για ε, το Μαυροβούνιο στο Κοινοβούλιο σε σχέση με άλλους οι οποίοι δεν έχουν τέτοια μακρά θητεία και παρόλα τα προβλήματα που μπορεί να υφίσανται σε σχέση με τον τουρισμό καμιά φορά και ίσως ε, και τα προβλήματα τα μεταναστευτικά με τις ροές μεταναστών μέσω των Δυτικών Βαλκανίων καταφέρατε να οδηγηθείτε σε μια αφούσα, σε μια ευημερούσα οικονομία παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σας. Αντιμετωπίζετε η διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα καταβάλλονται προσπάθειες και βρίσκεστε καθοδόν προς την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπούμε πρέπει να το πω ως μόνιμος συγητής μετά από 7 χρόνια και είναι μια προσωπική δήλωση που κάνω τώρα ακολουθώντας τη διαδικασία για το Brexit που είναι ιδιαίτερα θλιβερή υπόθεση εγώ ήμουν εναντίον της αποχώρησής μας θα είναι η τελευταία μου η έκθεση του Νοεμβρίου και με το άρθρο 50 που θα ξεκινήσει για την αποχώρηση ε, για την εφαρμογή του για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνω έκκληση σε εσά. παρακαλώ μην πιεστείτε σε σχέση με τα θέματα της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μην αποθηθείτε ε, λόγω του Brexit είναι πραγματικά πολύ απαιτητική η καιρή και μεγάλες οι προκλήσεις αλλά είναι επιθυμητή η ιδιότητα μέλους της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευελπιστώ θα συνεχίσετε με τις προσπάθειές σας να ενταθείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλη την απόφαση που έλεγα η δική μου χώρα να αποχωρήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ δόκτωρα Τένο και τις παρατηρήσεις σας. Συγκινούμε από τα όσα είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να το αναφέρω αυτό για την ε, συζήτηση για την, ε, το να γίνει κάποιος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά κεφάλαια σε σχέση με το Μαυροβούνιο, έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε σχέση με άλλες χώρες και αυτό πρέπει να το δηλώσουμε για να αποφευθούν παρεμηνίες. Και ο λόγος που εκφωνήθηκε χθε για την προπαρασκευή της Συνόδου της Μπρατισλάβας ώστε να ε, προετοιμαστεί η διαδικασία μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κάλυψε όλα τα θέματα επί του επιστητού να μην υπάρξουν παραμηνίες λοιπόν και λόγω αυτού σας ζητώ λοιπόν να είσαστε λίγο πιο σύντομοι στις παρεμβάσεις σας στη συζήτηση, γιατί στις 9 θα, ακριβώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε ακριβώς με το επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη. Και θα πρέπει να υπάρξει αρκετό χρόνο για να απαντήσει σε ερωτήσει ο Πρωθυπουργό Τζουκάνοβιτ. Ο κ. Σαμπάρα έχει τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι προνόμιο για μένα ως φιλελεύθερο ε, που επισκέφθηκα φέτος το καλοκαίρι τη χώρα σας ε, προσκεκλημένος του Ανδρέα Πόποτευστη. Ήταν η πρώτη μου επίσκεψη στη χώρα σας, η οποία ήταν, ε, βρήκα καλά οργανωμένη και αυτό είναι κοπλιμέντο για σας. Προχωρούν οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση καλά και τώρα ουσιαστικά είστε μέλος του ΝΑΤΟ. Το ερώτημά μου είναι, αυτό δεν αρέσει φυσικά στους Ρώσους, το γεγονός ότι είστε τόσο κοντά στη Δύση και τόσο μέσα στο ΝΑΤΟ. Σας ε, άσκησαν πιέσεις, σε εσάς ή στους συμπατριώτες σας, δηλαδή ποιες είναι οι σχέσεις της χώρας σας με τη Ρωσία. Thank you very much. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να σας καλωσορίσω εκ μέρους της ομάδας μου των Πρασίνων Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ. Θέλω να σας συγχαρώ όχι μόνο για τα 10 χρόνια της ανεξαρτησίας της χώρας σας, αλλά και για την προόδο που σημείωσε η χώρα σας κατά την ε, εφαρμογή του κεκτημένου. Όπως είπε και ο πρόεδρος της ομάδας μας, είστε, ε, του, της Επιτροπής μας, είσαστε μια χώρα που έχει προχωρήσει πολύ σε σχέση με την περιοχή σας. Και η, το Κοινοβούλιο στηρίζει πολύ την διαδικασία διεύρυνσης, τόσο η δική μου ομάδα αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία των παρισταμένων. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, επίσης σας συγχαίρω για το γεγονός ότι και εσείς και άλλοι στη χώρα σας ολοκληρώσατε τη διαδικασία μετάβασης προς εκλογές. Όπως είπε ο ε, εισηγητής, υπάρχει πλουραλισμός με μια κυβέρνηση ε, που περιλαμβάνει περισσότερες πλευρές και, και στο σε δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες θα έρθει ο νέος πρόεδρος του κοινοβουλίου σας, το κοινοβούλιο μας. Το κόμμα του ήταν πολύ σημαντικό στο να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία μετάβασης. Λοιπόν, σχετικά με αυτή τη διαδικασία, δύο ερωτήσεις. Μία από τις συμφωνίες ήταν ότι τα ψηφοδέλτια και οι εκλογικοί κατάλογοι, οι εκλογικοί κατάλογοι θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί. Ε, ακούω ότι δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία όσο θα έπρεπε. Είσαστε σίγουροι ότι μέχρι την ημέρα των εκλογών θα έχουν ενημερωθεί εκλογικοί κατάλογοι για να μην υπάρχουν προβλήματα κατά τις εκλογές. Δεύτερο ερώτημα που αφορά την περίοδο μετά τις εκλογές. Όσον αφορά την πολιτική σταθερότητα, πώς προβλέπετε ότι θα, ποια προβλέπετε θα είναι η πολιτική σκηνή, ποιοι θα είναι οι εταίροι σας στην κυβέρνηση και σχετικά με το ΝΑΤΟ. Πιστεύετε ότι όλοι οι συμμαχοί σας θα σας ε, υποστηρίξουν μετά τις εκλογές στην συμμετοχή σας στο ΝΑΤΟ τελευταία ερώτηση από πλευράς Πρασίνων σχετικά με την ε, οικοδόμηση του δεύτερου μέρους του θερμοδυναμικού ε, εργοστασίου στην Πλάβια. Από ό,τι ακούω αυτό δεν ε, συμφωνεί με τη Συμφωνία των Παρισίων για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Πώς θα τα καταφέρετε αυτά εσείς ως υπό ένταξη χώρα πρέπει να κάνετε ό,τι κάνουν και οι άλλες ε, χώρες, μέλη της Ένωσης ή οι υποψήφιες χώρες για να λειτουργήσει η διαδικασία των Παρισίων. Λοιπόν, ε, τι συμβαίνει εδώ, γιατί ακούω ότι δεν συμμορφώνεται απόλυτα αυτή η μονάδα. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, σας ε, καλωσορίζω και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ήθελα να σας ρωτήσω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, υπογράψατε συμφωνία με τον ΝΑΤΟ από ποιε απειλέ θεωρείτε ότι θα προστατεύσει τη χώρα σας στο ΝΑΤΟ. Και δεύτερη ερώτηση, με ποια στοιχεία της νέας στρατηγική του ΝΑΤΟ συμφωνείτε και πώς περιμένετε να τα εκμεταλλευτείτε αυτά προς το συμφέρον της χώρας σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να ξεκινήσω με τρει φορέ συγχαρητήρια, τριπλά συγχαρητήρια. Πρώτον, για την δέκατη επέτειο τη ανεξαρτησία τη χώρα σα, σα συγχαίρω. Δεύτερον, σα συγχαίρω για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί για να γίνετε κράτος μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, σα συγχαίρω για τι προσπάθειε τη ένταξη με τον ΝΑΤΟ. Δεν έχω συγκεκριμένη ερώτηση. Συμφωνώ μαζί σας όταν κάνετε λόγο για τη σπουδαιότητα της ειρήνης και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή σας. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οι πηγές πιθανών σειράξεων και τριβών δεν έχουν καταργηθεί, δεν έχουν αρθεί και μάλιστα σε μονιμότερο πλαίσιο. Γίνεται λόγος για εξελίξεις και ανάπτυξη. Ανάπτυξη προς όφελος ευρύτερα της Ευρώπης και εσείς ως πολιτικός γνωρίζετε σίγουρα ε, προς ε, γίνεται αυτή η αναφορά για την Ευρώπη και για το ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ σημαντική η στάση και της κυβέρνησής σας και των άλλων πολιτικών δυνάμεων στο Μαυροβούνιο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία για ευτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you, Mr. Chair. Uh, from the group, from the social... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και από του σοσιαλδημοκράτες και εμείς θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για τα 10 χρόνια ανεξαρτησία της χώρας σας και όπω είπε και ο κύριο Μπρόκ με επιτυχή τρόπο ολόκληρο προχωράτε. Έχετε ανοίξει 24 κεφάλαια μέχρι σήμερα και ευχόμαστε να ολοκληρώσετε και με τον ταχύτερο κιόλας τρόπο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει έντονο το αίσθημα ότι οι διαδικασίες ένταξης του Μοντενέγκρο θα στεφθούν με επιτυχία για να γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης καλή επιτυχία στις για τις επικείμενες εκλογές και ευελπιστούμε ότι θα ανταποκρίνονται οι προδιαγραφές σε σχέση με τις εκλογές που θα διεξαχθούν με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Δύο ερωτήσεις έχω. Είναι οι εξή. Γίνεται επίσης λόγο για τις άλλες χώρες και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα των προτεραιοτήτων. Ποιε είναι οι προτεραιότητε τη κυβέρνησή σα για να καταπολεμηθεί η διαφθορά που είναι ένα πρόβλημα για όλου Καταπολέμηση λοιπόν της διαφθοράς, ε, διασφάλιση όρων και προϋποθέσεων που είναι ακρογωνίως λίθος ε, αυτό το ζήτημα για ε, την προσέγγιση σας στην Ευρώπη. Επίσης είδαμε και να αναδύεται ο εθνικισμός και πάλι στην περιοχή σας. Εθνικιστικές εξάσεις με το πιο πρόσφατο παράδειγμα τις διαδηλώσεις, ε, την αντίσταση σε σχέση με το κοσυφοπέδιο όσον αφορά την, τον καθορισμό συνοριακών γραμμών στις πρόσφατες εξελίξεις. Ποια είναι η στάση σας σε σχέση με αυτή την κατάσταση, ποιες είναι οι προοπτικές, πώς τις βλέπετε. Σας ευχαριστώ, κάθε επιτυχία ευχόμεθα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε θετική απήχηση και σας ευχαριστούμε για τα θετικά μηνύματα όταν λέτε ότι είσαστε πρόθυμος και έτοιμος να συνεχίσετε να δώσετε συνέχεια στη διαδικασία προσέγγισης δράποσμο Αληθεύει ότι εχθές ο κύριος Γιούγκερ δεν ανέφερε συγκεκριμένα με, εξειδικευμένο τρόπο τη διαδικασία διεύρυνσης μεταξύ των προτεραιοτήτων του. Αληθεύει όμω ότι στον, εξωτερικό, στον εξαιρετικό λόγο που εξεφώνησε δεν ανέφερε και άλλα σημαντικά θέματα όπως τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας ή τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. έχω την ακράδαντη πεποίθηση ότι λοιπόν η διεύρυνση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παραμένει προτεραιότητα στον πρώτο γύρο για τον κύριο Γιούγκερ και την Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης να πω ότι κατά την προηγούμενη θητεία σας είσαστε υπέρμαχος, είχατε έναν υπέρμαχο τον κύριο Τάνοκ ως εισηγητή για το Μαυροβούνιο. Θλίβομαι που θα αποχωρήσει πλέον από αυτό το αξίωμα. Υπάρχει όμως η βεβαιότητα ότι έχετε πάρα πολλούς φίλους στο, για ε, το Μαυροβούνιο σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Σε σχέση με την άνοδο του εθνικισμού και τις τριβές ε, σε σχέση με το παρελθόν στα Βαλκάνια, τι πιστεύετε ότι μπορείτε εσείς να κάνετε για να σβήσει αυτή η φωτιά, να πάψουν αυτά τα προβλήματα και οι τριβές. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Μια και θα πρέπει να αποχωρήσω τώρα. Θα ήθελα να παρακαλέσω ο συνάδελφος Πλένκοβιτς να αναλάβει την προεδρία τη συνεδρίασής μας. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω εσάς για την πολύ καλή συνεργασία, αντικειμενική και δημιουργική συνεργασία που είχαμε κατά το τελευταίο διάστημα εδώ. Είναι καλό να το ξέρει κανείς ότι μπορεί να έχει έναν έμπιστο εκπρόσωπο, τίποτα δεν μπορεί να πάει έτσι στραβά. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την εκλογή σου στην Κροατία και τα όσα θα απορρέψουν από αυτήν. Έχετε λοιπόν την προεδρία. Και πραγματικά καλό είναι το ότι εσύ θα ηγηθεί στι συνεδρίε αυτή, διότι γνωρίζουμε ότι στα Βαλκάνια υπάρχουν πολλέ εντάσει από το παρελθόν και πολλά προβλήματα δεν έχουν ακόμα διευθετηθεί, δεν έχουν επιληθεί. Είναι αναγκαίο να υπάρξουν ηγέτε αυθεντική ηγεσία στα Βαλκάνια με ευρωπαϊκές πρόπτικες και κατευθύνσεις. Η Ευρώπη τα σύνορα τα καθιστά περιτά δεν τα καταργεί αλλά τα καθιστά περιτά και έτσι πολλά προβλήματα καθίστανται πιο εύκολα επιλύσιμα υπό αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα. Α σκεφτεί κανεί τη σχέση μεταξύ Γερμανία και Γαλλία. γι' αυτό σας εύχομαι κάθε επιτυχία σε εσά ώστε στη διαδικασία αυτή ευρύτερα στα Δυτικά Βαλκάνια να στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια σε σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Παρακαλώ να αναλάβετε την Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ, Έλμαρ Μπροκ. Τώρα ο Εντουάρτ Κούκαν παρακαλώ θα λάβει τον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ΑΦΕΤ. Ε, είναι πάντοτε ευχαρίστηση να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με έμπειρους πολιτικούς ε, όπως εσείς. Σας ε, συγχαίρω επίσης και για τη δέκατη επέτειο της ανεξαρτησίας σας. Όπως γνωρίζετε η Σλοβακία ήταν πολύ ένθερμα παρούσα όταν γεννήθηκε το ανεξάρτητο Μαυροβούνιο. Πάντοτε προσπαθούμε να βοηθήσουμε ως ε, χώρα προεδρίας θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε το κλείσιμο κεφαλαίων, ενταξιακών κεφαλαίων. Ο κύριος Μπρόκ, ο πρόεδρος μας, είπε ότι είστε ε, πρωτοπόρος της περιοχής στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό θα διαπιστωθεί και θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Δύο πράγματα ε, θέλω να πω σε σχέση με τη θέση σας. Υπάρχουν προβλήματα, υπήρξαν προβλήματα την προηγούμενη δεκαετία. Κανείς όμως δεν μπορεί να αρνηθεί τις μεγάλες επιτυχίες του Μαυροβουνίου στην πορεία. Σύντομα θα είμαστε εταίροι στα πλαίσια της βορειοατλαντικής χυσίας. Και όσον αφορά τη διαδικασία της διεύρυνσης, εκτιμάμε ότι έχετε πλήρως συνταχθεί με την CFSC ε, στις δύσκολες αυτές συνθήκες. Αυτό είναι πολύ θετικό. Όπως επίσης η δέσμευσή σας ε, η εμπλοκή σας με άλλες χώρες της περιοχής, η καλλιέργεια καλών σχέσεων είναι πάντοτε σημαντική. Όσον αφορά τις εκλογές, κύριε Πρωθυπουργέ, θα γίνουν τον Οκτώβριο στα πλαίσια ενός νέου νόμου, θα είναι ένα μια ε, ε, δοκιμή για το αν θα έχουν ληφθεί υπόψη οι συστάσεις του ΟΝΤΙΡ. Και το ερώτημά μου είναι πώς αισθάνεστε εν ώψη αυτών των εκλογών. Και ευχαριστώ πολύ, Εντουάρντ κύριος Ευχαριστώ. Καλωσορίζετε ορίσατε στο Στρασβούργο, κύριε Πρωθυπουργέ. Θέλω να σας συγχαρώ και εγώ για την δέκατη επέτειο τη ανεξαρτησία σας. Ως ε, εισηγητής των σοσιαλιστών για την Βοσνία ε, Ερζεγοβίνη, ανησυχώ για τις εξελίξει εκεί, κυρίως στη Ρεπούμπλικα Σέρφκα το Μαυροβούνιο κατάφερε να προχωρήσει με επιτυχία προς την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Επίσης, οι σχέσεις ε, Μαυροβουνίων και Βοσνίων έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Είστε, έχετε φιλικές σχέσεις με όλους τους εμπλεκόμενους στην πολιτική ζωή της Βοσνίας υπάρχει η οργάνωση των ε, κοινωνιών, της οργάνωσης των κοινωνιών μετά τις ε, συγκρούσεις. Ποια είναι η γνώμη σας από αυτού. Ευχαριστώ τώρα, το λόγο έχει ο Πέτρος Οστροβίτσιος. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε απόλυτο δίκιο. Ένας τρόπος μόνο υπάρχει να χτιστεί το μελλοντικό ε, μαυροβόνιο, οι πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Εγώ υπήρξα επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας μου, το ξέρω, το ξέρω από την εμπειρία μου λοιπόν, ποια αποτελέσματα πετύχαμε. Ήδη έχετε την εμπειρία του, της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Όταν είδαμε τις διαδηλώσεις που οργανώθηκαν στη χώρα σας κατά της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Θέλω να σας ρωτήσω για την ε, υποστήριξη, της, για την διάθεση της κοινή γνώμης ε, την ένταξη στην ομάδα των δυτικών πολιτισμένων χωρών όπου υπάρχει κράτος δικαίου. Ε, πόσο χρόνο αφιερώνετε στο να εξηγείτε στην κοινή γνώμη όλα αυτά τα θέματα γιατί η υποστήριξη από την κοινή γνώμη είναι καθοριστική σημασίας για την πραγματική ένταξη στην ομάδα ανθρώπων που έχουν τις ίδιες απόψεις και είστε φυσικά πολύ ευπρόσδεκτοι σε αυτή. Ευχαριστώ η Σάντρα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, βρίσκομαι εδώ, εδώ, εδώ δεξιά σας όπως και ο Πέτρας ε, ε, προέρχομαι από τις χώρες της Βαλτικής. Γνωρίζω τι θα πει να είναι κανείς χώρα υποψήφια και να που διαπραγματεύεται την ένταξή της. Γι' αυτό θέλω να σας συγχαρώ για τη σημαντική προόδο του Μαυροβουνίου στην πορεία των διαπραγματεύσεων για ένταξη. Όπως επίσης και για τα, αυτά που πετύχατε για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Είναι μια πολύ σημαντική ένδειξη η ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ε, ε ένα σημάδι προς ε, την ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Ε, λυπάμαι που οι δεσμεύσει της ε, Θεσσαλονίκης ότι υπάρχει ευρωπαϊκό μέλλον για τα Δυτικά Βαλκάνια εφαρμόζεται πάρα πολύ αργά για δυσκολίες και, λόγω δυσκολιών και από τις δύο πλευρές. Και επίσης λυπάμαι που ο ενθουσιασμός για τη διεύρυνση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αρχίσει να μειώνεται. Παρά τα αυτά έγινε, απόφαση το Big Bang το 2004. Γνωρίζω ότι η κρίση στο χωσιφοπαίδιο έδειξε στους Ευρωπαίους πόσο σημαντική είναι η σταθεροποίηση της περιοχής. Πιστεύω επίσης ότι και η μεταναστευτική κρίση θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους να κατανοήσουν ότι δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε την αποσταθεροποίηση της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. Σας εύχομαι επιτυχία στις εκλογές. Είναι σημαντικό το αποτέλεσμα να δώσει κυβέρνηση που θα ασχολείται με τις μεταρρυθμίσεις και θα συνεχίζει την πλήρη υποστήριξή της προς την ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σάντρα. Εξαντλήθηκε ο κατάλογος των ομιλητών. Ήμουν και εγώ στον ε, κατάλογο. Παίρνω το λόγο. Ε, με τις ευκαιρίες αυτές που υπάρχουν Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τον γρήγορο ρυθμό τον οποίο ακολουθείτε για την ε, ένταξή σας στην ευρωπαϊκή οικογένεια όπως επίσης και για την ένταξή σας ε, στο ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι με το ρυθμό αυτό και παρά τις ε, αλλαγές κλίματος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από το θέμα ε, της διεύρυνσης, εσείς θα συνεχίσετε στον σωστό δρόμο. Σας συγχαίρω λοιπόν εξ ονόματος και της Κροατίας και θα κάνω ό,τι μπορώ έτσι ώστε οι διμερείς σχέσεις ε, να προωθηθούν, τα προβλήματα να λυθούν στα πλαίσια του πνεύματος ευρωπαϊκής συνεργασίας. Είναι σημαντικό αυτό για την περιοχή μας. Έχετε το λόγο κύριε Πρωθυπουργέ και έχετε το πολύ 10 λεπτά για να δώσετε απάντηση στις ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πλέκοβιτς. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για την υποστήριξη την οποία έχετε εκφράσει μέχρι σήμερα. Θέλω λοιπόν για μια ακόμη φορά κύριε Πλάνκοβιτς να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ πριν από οτιδήποτε άλλο για τα εξαιρετικά αποτελέσματα στις εκλογές στην χώρα σας. Ελπίζω γρήγορα να σχηματίσετε την κυβέρνησή σας η οποία είμαι σίγουρος ότι θα προωθήσει και τις καλές σχέσεις γειτονίας. Ε, θα είμαι σύντομος. Ακούστηκαν κάποια σχόλια για κάποιες εναλλαγές ύφους από πλευράς Βρυξελών σε σχέση με το θέμα της διεύρυνσης γενικότερα. Ε, εγώ θα ήθελα να ακούσω, είναι αλήθεια, μια πιο ενθαρρυντική αν θέλετε ε, κατάσταση από πλευράς των Βρυξελών. Πάντως, Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι οι Βρυξέλλες ε, να κατανοήσουν ακριβώς τις επιπτώσεις ε, της νέας κατάστασης που δημιουργείται για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης ε, της περιοχής μου. Τώρα γενικότερα για την περιοχή μου, για τα Δυτικά Βαλκάνια, <coughs> νομίζω ότι μέσω της ευρωπαϊκής πορείας μέσω της λεγόμενης πορείας του Βερολίνου, της διαδικασίας του Βερολίνου, έχουμε προσθέσει μια νέα διάσταση στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εμείνουμε προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να βελτιώσουμε και να ενημερώσουμε σε εισαγωγικά την ίδια τη διαδικασία του Βερολίνου, γιατί νομίζω έτσι θα βοηθηθούν οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Ευχαριστώ τους εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εμπλοκή τους στις διαδικασίες αυτές. Τους ευχαριστώ πολύ. Και να πω ότι η νέα κυβέρνηση θα συνεισφέρει στην πολιτική σταθεροποίηση της χώρας μου και θα επιτρέψει τις δυνάμεις της χώρας μου να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στα θέματα της οικονομικής ανάπτυξης με πλήρη σεβασμό των δημοκρατικών διαδικασιών και των δικαιωμάτων των πολιτών. Έτσι και οι πολίτες της, ε, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου ε, αποφάσισαν κάτι το οποίο είναι σεβαστό εμείς στο ε, Μαυροβούνιο ε, μένουμε στα την Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζουμε ότι μέσω της συνέχισης των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών θα συνεισφέρουμε γενικότερα στην υπόθεση της Ευρώπης. Αναφερθήκατε στις θέσεις της αντιπολίτευσης σε σχέση με το πιθανότητα δημοψηφίσματος για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Ε, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι μια πρωτοβουλία θα έλεγα των κομμάτων αυτών. Ξέρετε ποιοι στην διεθνή κοινότητα είναι υπέρ ενός τέτοιου δημοψηφίσματος διότι ελπίζουν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να καθυστερήσει ε, τη χώρα μου να γίνει ε, μέλος του ΝΑΤΟ και φυσικά η αντιπολίτευση η οποία επιθυμεί να αναλάβει την εξουσία χρησιμοποιεί κάθε τέτοια στάση αν θέλετε και προσπάθεια έτσι ώστε να έχει η ίδια ε, την δυνατότητα να κερδίσει. Ε, εγώ θα ήθελα να πω ότι το σύνταγμα της ε, χώρας μου δεν καθιστά ένα τέτοιου είδους δημοψήφισμα υποχρεωτικό. Αν το κοινοβούλιο της χώρας πάρει μια τέτοια απόφαση, τότε σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε. Αλλά νομίζω ότι είναι το κοινοβούλιο κυρίαρχο να αποφασίσει για το τι θα γίνει. Εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω το τι θα αποφασίσει το επόμενο κοινοβούλιο, διότι θα έχουμε πολύ σύντομα εκλογές. Είμαι βέβαιος όμως ότι το δικό μου κόμμα μετά τα αποτελέσματα ε, θα παραμείνει ένα σημαντικός παίκτη ε, ε, ε, στο παιχνίδι της εξουσίας στο Μαυροβούνιο και θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει. Πάντως επαναλαμβάνω για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, το νέο κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο θα πάρει τις αποφάσεις οι οποίες απαιτούνται να ληφθούν. Το ότι η Ρωσία δεν της αρέσει το ότι κοντά στο ΝΑΤΟ και μας κάνατε ερωτήσεις για τις σχέσεις μας ουσιαστικά με τη Ρωσία. Θα ήθελα να πω ότι στην ιστορία η Ρωσία και το Μαυροβούνιο έχουν πολύ στενές σχέσεις. Έχουμε γιορτάσει πρόσφατα αιώνες στενών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό δεν είναι όμως κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει στο να αποκλίνουμε από την βασική μας προοπτική που είναι η υιοθέτηση ενός νέου συνόλου αξιών που θα μας οδηγήσει στην πλήρη ένταξη της, ε, ε, στις ε, στην ολοκλήρωση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό δεν θα πρέπει να κλονίσει τις σχέσεις μας με αυτούς τους παλαιούς φίλους. Δεν το κάνουμε εμεί σε καμία περίπτωση για να υπονομεύσουμε τις παλαιές παραδοσιακές μας σχέσεις. Εμείς απλά επιδιώκουμε να εξυπηρετήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Έχουμε επιλέξει να γίνουμε μέρος της ευρωατλαντικής κοινότητας. Αυτή είναι η πολιτική μας. Τώρα, αυτό δεν αρέσει στη Ρωσία. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν τους αρέσει αυτό γιατί πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο θα επηρεάσει γενικότερα τις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Ε, ελπίζω ότι οι σχέσεις αυτές που δεν είναι καλές σήμερα να βελτιωθούν στο μέλλον. Πριν μερικά χρόνια οι σχέσεις δεν ήταν κακές. Ε, τον τελευταίο καιρό έχουν ε, κατά κάποιο τρόπο επιδεινωθεί. Πάντως νομίζω ότι θα υπάρξει ε, μια επιτυχής κατάληξη των προσπαθειών μας να διαβεβαιώσω την κυρία Λούνατσεκ ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να ενημερωθούν οι εκλογικοί κατάλογοι με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, με όλους τους εμπειρογνώμονες ε, οι οποίοι απαιτείται να βοηθήσουν. Ένα λάθος είχε γίνει στο παρελθόν το οποίο ελπίζουμε ότι θα διορθώσουμε. Είναι όμως σαφές ότι από εδώ και πέρα ε, είμαστε σε θέση να διασφανίσουμε ε, την κανονικότητα των εκλογικών διαδικασιών. Τώρα τι κυβέρνηση θα είναι η επόμενη κυβέρνηση στη χώρα μου. Ε, αν η κυβέρνηση αυτή θα εμείνει στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Ναι, νομίζω ότι ναι θα εμείνουμε στην ένταξή μας στην Ευρώπη, θα εμείνουμε στην πορεία μας προς τις ε, ε, νατοικές δομές. Νομίζω ότι η νέα κυβέρνηση θα είναι σε θέση να συγκεντρώσει την προσοχή της στις βασικές προτεραιότητες τις οποίες έχουμε στην εξωτερική πολιτική. Ε, για την μονάδα παραγωγής ενέργειας της Πλάβια, Νομίζω ότι όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας αποδεικνύουν ότι σεβόμεθα πλήρως τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών σε διοξίδιο του άνθρακα. Και ο Έλλην φίλων μας είπε τι απειλές είναι αυτές από, τα, από τις οποίες θα κληθεί η Ρωσία να μας προστα... η... το ΝΑΤΟ να μας προστατεύσει. Κοιτάξτε, ε, δεν είναι άμεσες απειλές δικές μας. Εμείς έχουμε όμως κάποια θέματα. Η περιοχή αυτή, είτε μας αρέσει είτε όχι, χαρακτηρίζεται από κάτι που θα ονόμαζα μόνιμη αστάθεια τον τελευταίο καιρό. Και η ιστορία έχει αποδείξει ότι από μόνοι μας ίσως θα είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα στο μέλλον. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι δικό μας, δεν έχουμε ένα ειδικό πρόβλημα εμείς. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε σε περιφερειακή ολοκλήρωση, σε ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Νομίζω ότι τα Βαλκάνια είναι τμήμα της Ευρώπης, ε, παραδοσιακά, πολιτισμικά ήταν σημαντικό κομμάτι της Ευρώπης και τελικά ε, εμείς σήμερα έχουμε καταλήξει να ε, είμαστε μια σημαντική οικονομία της περιοχής έχουμε όμως ένα χαμηλό τελικά κατακεφαλήν εισόδημα πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας προσπάθεια για να ανακτήσουμε αν θέλετε ε, τις διαφορές αυτές, για να καλύψουμε καλύτερα τις διαφορές αυτές και αυτό θα ανοίξει νέες δυνατότητες ε, και στον οικονομικό τομέα. Για τον κύριο Πέτερλε σας ευχαριστώ επίσης για τα καλά σας λόγια, για την υποστήριξή σας προς την χώρα μου. Θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπατε ότι εξακολουθούν όπως είπα να υπάρχουν πηγές ε, περιφερειακής αστάθειας. Βλέπουμε τι έγινε και τον τελευταίο χρόνο. Ε, σε κάποιες ε, περιπτώσεις στο παρελθόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση οι προοπτικές μας παραμένουν καλές όμως ταυτόχρονα υπάρχουν και ορισμένα μηνύματα. Μηνύματα που λαμβάνονται ότι δηλαδή οι πηγές ε, αστάθειας ε, εξακολουθούν να υφίστανται και νομίζω ότι συμφωνούμε αμφωτέρωθεν ότι πρέπει να προαγάγουμε, να δώσουμε μια νέα όθηση στις προσπάθειες ε, ολοκλήρωσης η ερώτηση που τέθηκε για τις προτεραιότητες της κυβερνητικές σε σχέση με την καταπολέμηση της διαφθοράς ε, αλλάξαμε, τροποποιήσαμε το νομοθετικό πλαίσιο στο Μαυροβούνιο. Έχουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο τώρα και νομίζω ότι σε σχέση με τα αποτελέσματα έχω ήδη κάνει λόγο για κάποια από αυτά. Πολλές προσπάθειες καταβάλουμε για να ε, μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, συστημικές ε, μορφές τέτοιου είδους ε, γεγονότων και πράξεων ώστε να μην συνεχιστεί η διαφθορά. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να απαλείψουμε από την εκπαίδευση, από την ε, περίθαλψη αυτά τα σημεία τα οποία μπορούν ίσως να δημιουργήσουν αιτίες και πηγές διαφθοράς. Όσον αφορά την άνοδο του εθνικισμού στην περιφέρειά μας και τις σχέσεις με το ποσυφοπαίδιο θα ήθελα να αναφέρω ότι εξακολουθούμε να δεσμευόμεθα όσον αφορά την ανεκτικότητα και την ενδυνάμωση και ε, αποτελεσματικότητα της ανεκτικότητας μεταξύ των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων και θρησκευτικών ομάδων. Το αποδείξαμε νομίζω έμπρακτα αυτό και τα αποτελέσματα ε, αποδείχθηκαν και στο υψηλό επίπεδο συνεργασίας με τους γείτονές μας. Δεν υφίστανται προβλήματα σε σχέση με τα σύνορα του Κωσυφοπεδίου όπως είχε συμβεί ε, με την Βοσνία Εζεγοβίνη. Υπήρξε για μια σύντομη περίοδο ένα πρόβλημα με τη Βοσνία Εζεγοβίνη. Ωστόσο αυτό οφειλόταν σε κυριότερα σε εσωτερική πολιτική κατάσταση που είχε προκαλέσει αυτή την, αυτό το αποτέλεσμα όταν υπήρξε μια πρωτοβουλία που ανελήφθη εκεί για την αλλαγή των συνόρων. Πολύ σύντομα μας αντελήφθησαν ότι οι συστάσεις ε, της Μπαντεντέρ, Επιτροπής Μπαντεντέρ της ε, δεκαετίας του 1990 για την μη τροποποίηση συνόρων που έπρεπε, ότι έπρεπε αυτές οι συστάσεις να είναι σεβαστές Έκτοτε δεν είναι προβλήματα. Δεν έχουμε και προβλήματα ούτε και με το κοσυφοπέδιο. Καμιά φορά υφίστανται προβλήματα όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές τριβές και συζητήσεις και τους διχασμούς εσωτερικά στο κοσυφοπέδιο. Έχει όμως αποσταλεί μήνυμα προς το κοσυφοπέδιο ότι είμαστε πρόθυμοι να υπογράψουμε και να επικυρώσουμε τη συμφωνία που υπεγράφει στη Βιέννη πριν από ένα έτος. Ε, όταν θα είναι έτοιμο λοιπόν το κοσυφοπέδιο θα υπογράψουμε και εμείς τη διακρατική αυτή συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούχαν ε, για τα λόγια σας που μας υποστηρίζετε και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δική σας συνεισφορά όσον αφορά τις παρεμβάσεις σας ε, υπέρ του Μαυροβουνίου για την ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως προοπτική του. Και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ κατά τα άλλα με αυτά τα οποία αναφέρατε για τη σπουδαιότητα της δέσμευσης του Μαυροβουνίου για καλές γειτονικές σχέσεις ε, με τα όμορα κράτη. Και συμφωνώ επίσης ότι οι επικείμενες εκλογές θα έχουν μεγάλη σπουδαιότητα, θα είναι μεγάλη εμβέλεια εκλογές. Ε, θα είναι μια επανεπιβεβαίωση όλων όσων έχουν ήδη γίνει κατά τα τελευταία αυτά δέκα χρόνια και των πρωτοβουλειών που ανα... ανα... είχαμε αναλάβει υπάρχει και μία μειονότητα αρκετά ισχυρή ωστόσο στα Δυτικά Βαλκάνια που εξακολουθεί να επιθυμεί να παραμείνει εκτός της διαδικασίας ολοκλήρωσης και ευρωπαϊκής προοπτικής. Εξακολουθεί λοιπόν να υφίσταται αντίσταση αυτών των μειονοτικών δυνάμεων. Σε άλλες χώρες όταν υπάρχει μια κυβερνητική αλλαγή πολύ συχνά εξακολουθεί η ίδια πολιτική να ακολουθείτε πολιτικά. Εδώ όμως ε, δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο αν υπήρχε κυβερνητική αλλαγή. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικές αυτές οι εκλογές. Υπήρξε και ερώτηση για το πώς θα μπορούσαν να επιληθούν ε, τα προβλήματα όσον αφορά την θρησκευτική ανεκτικότητα την ανεξιθρησκεία. Το ανέφερα αυτό. Έχουμε πολυετή παράδοση ε, στη χώρα μας σχετικά. Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια, ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να βελτιώσουμε περαιτέρω αυτή την ήδη θετική κατάσταση. Είναι ένα πολύ θετικό παράδειγμα, ένα υπόδειγμα το Μαυροβούνιο ως προς αυτά και στο Μαυροβούνιο οι μειονότητες όλες οι μειονότητες υποστήριξαν την πρωτοβουλία που είχαμε αναλάβει για να κερδίσουμε την ανεξαρτησία μας αποστέλλοντας ένα σαφέστατο μήνυμα ότι πίστευαν σε αυτή την ανεξαρτησία και επιθυμούσαν να υπάρξει η ευθύνη που θα αναλαμβάναμε της κρατικής υπόστασης και ανεξαρτησίας μας και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό Επίσης, ευχαριστώ για τις πολύ θετικές συμβουλές που μας δώσατε με βάση την μεγάλη πείρα σας και όταν έχουμε θέματα δημόσιας ε, της διάθεσης των πολιτών μας ε, και πώς αντιμετωπίζεται η τάση έντασης ή η ένταξη στο ΝΑΤΟ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια αύξουσα τάση ε, υπέρ αυτής της προσπάθειας. Ό,τι κάνουμε ε, για, την, ε, ε, να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πολιτική μας Α, όλα αυτά μας επιτρέπουν να σημειώνεται ένα μεγάλο ποσοστό υποστήριξης υπέρ, της, υπέρ του ΝΑΤΟ. Πέρα από όλα αυτά μπορώ να σας πω ότι όλες οι σφιγμομετρήσεις και τα βαρόμετρα δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών γνωρίζει ότι θα είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ το Μαυροβούνιο και οποιαδήποτε είναι η δική τους στάση ή θέση δεν θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτή την προοπτική, με αυτή την κατάσταση. Δεχθήκαμε συγχαρητήρια και <clears throat> όσον αφορά την συμφωνία της, του θεματολογίου της Θεσσαλονίκης και πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με όλα αυτά η όθηση για την περιφερειακή ολοκλήρωση και την ε, ε, ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρή όσο θα έπρεπε, αλλά υφίσταται όμως αυτή η τάση και αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ και, σας, και συμφωνώ με όσα είπατε για την κρίση στο Κωσίφο Πέδιο. Η κρίση του 1999 ήταν μια σημαντική προειδοποιητική βολή όσον αφορά τους άμεσα εμπλεκόμενους ε, έτυχε μεγαλύτερης προσοχής η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και πιστεύω ότι και η μεταναστευτική κρίση θα έχει πάλι την ίδια, τις ίδιες συνέπειες. Αυτές είναι προτεραιότητες όχι μόνο της ΕΕ αλλά και της δικής μας χώρας. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε να αναφερθεί ότι η διαδικασία διεύρυνσης θα έπρεπε να εξεταστεί ως μια πιθανή λύση Φυσικά τα προβλήματα της Ευρώπης, τα προβλήματα στην Ευρώπη και η ίδια η κρίση μας αποκαλύπτουν, μας δείχνουν κάποια αρχιτεκτονικά προβλήματα που υφίστανται στην δομή της Ευρώπης. Όμως αυτό δεν αποτελεί λόγο να εγκαταληφθεί η προσπάθεια και θα πρέπει να συνεχιστεί η, το να τονίζουμε την αξία αυτών των αξιών. Σας ευχαριστώ. Napravit ćemo malu pauzu prije nego što nam se priključi. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν, εύχομαι σε όλους ό,τι kalitero και θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα περιμένοντας τον Δαλάι Λάμα. Nathalie Nathalie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

Bitte Platz zu nehmen. Παρακαλώ καθίστε. Είναι πολύ Σας ευχαριστώ Δαλάι Λάμα που ήρθατε σε μας ε, σήμερα. Δεύτερη φορά από το 2006 που προσέρχεστε στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και πάλι εκ νέου για το ότι βρήκατε τη δυνατότητα να προσέλθετε σε εμά. Και πιο πριν υπήρξε και μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και πρέπει να μεριμνήσουμε και να δούμε ότι αυτές οι συζητήσεις πραγματικά, μια και είναι τόσο σημαντικές για μας, πρέπει να διεξάγονται. Είναι ένας μεγάλος θρησκευτικό ηγέτης θεωρούμε ο Νταλάη Λάμα και σε μια περίοδο πολέμων και βίας το μήνυμά του για τη μία άσκηση βίας με βάση αξίες και αρχές είναι για μας πραγματικά αδιάφορο σε ποια πίστη ανήκει κανείς για μας το μήνυμα αυτό είναι τεράστια σημασίας γι' αυτό πραγματικά δημονούμε να ακούσουμε τι θα μας πείτε και πραγματικά είναι απόλυτα σαφές ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε υπέρ της One China Policy μιας Κίνας, πολιτική μιας Κίνας. Δεν ζητάμε με κανένα τρόπο τον κατακαιρματισμό της Κίνας και δεν υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο. Και αυτή ήταν πάντα και η πολιτική του Δαλάη Λάμα, δηλαδή το θέμα της ε, αυτονομίας ε, για το θηβετιανό λαό πάντα τίθεται στο πλαίσιο αυτό, ώστε οι θρησκευτικές αξίες να μπορούν να ανθίσουν σε σχέση με το θηβετιανό λαό στο Θιβέτ, είναι μια απέτηση κάθε ομολογίας, κάθε θρησκείας, κάθε εθνικότητας να υφίσταται αυτό το δικαίωμα ώστε θρησκευτικές ταυτότητες και πολιτιστικές ταυτότητες να μην χάνονται, να μην διαλύονται. Και πρέπει να δούμε ότι και αυτό το οποίο είναι τεράστια σημασία, δηλαδή αυτό που στην Ευρωβουλή είναι το θέμα των κλιματικών αλλαγών που μας απασχολεί συχνά, στο οροπέδιο υψίπεδο του Θιβέτ που είναι μια ξεχωριστή περιοχή με τεράστια σημασία παγκόσμια και αυτό πρέπει να ενταχθεί λοιπόν. Δεν στρέφεται εναντίον κανενός αυτή η προσπάθεια και πρέπει να μπορούμε να συζητούμε ο ένας με τον άλλο για να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο κόσμο. Και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που η αγιότητά σας είσαστε εδώ ανάμεσά μας και μπορέσατε να προσέλθετε. Έχετε αμέσως τον λόγο. Παρακαλώ. Respected brother. Σεβαστοί αδερφοί και αδερφές, πάντοτε σας περιγράφω ως ανθρώπους, χωρίς διαφορές. 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι που ανήκουμε στην οικογένεια του ανθρώπου. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, αισθάνομαι μεγάλη τιμή που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Είμαι θαυμαστής του πνεύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. το δικό μας πρόβλημα στο, Θιβέ, στο Θιβέτ είναι κάτι που το συσχετίζω με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν θέλουμε να διαχωριστούμε από το λαό της Κίνας. Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά μας, βλέπετε. Δεν επιδιώκουμε ανεξαρτησία. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε υπέρ του διαχωρισμού, όμως δεν είμαστε υπέρ της απόσχησης. Όμως η κινέζικη ηγεσία αναφέρεται συνέχεια σε αυτό, στην απόσχηση. Όσον αφορά την πολιτική ευθύνη για το Θιβέτ, από το 2011 ήδη αποσύρθηκα εντελώς. Τα θέματα πλέον αυτά τα χειρίζεται μια εκλεγμένη πολιτική ηγεσία. Εγώ πλέον είμαι μεγάλος ηλικία, 81 ετών. Κοιτάξτε με όμως μοιάζομαι 81 ή μήπως σας φαίνομαι νεότερος. Έτσι λοιπόν, μόλις τώρα ο φίλος μου μου είπε «Ποιο είναι το μυστικό σου» και φαίνεσαι τόσο νέος. Και φυσικά πάντοτε εγώ απαντώ, αυτό είναι μυστικό, δεν το αποκαλύπτω. Όμως, έχω εκπαιδεύσει το νου μου, το μυαλό μου, με έναν τρόπο που εφαρμόζω αυτό που ονομάζουμε αναλυτικό διαλογισμό. Και με αυτό τον τρόπο λειτουργεί το μυαλό μου. Πολλές πολλά καταστροφικά συναισθήματα, όπως η οργή και ο φόβος, δεν έχουν λόγο να υπάρχουν. Με πραγματική ανάλυση μπορεί κανείς να προχωρήσει με τη συμπόνια. Και αυτό υποστηρίζεται και από επιστημονικές έρευνες. Αυτό είναι λοιπόν το μυστικό μου. Όλοι έχουμε τις ίδιες δυνατότητες να γνωρίζετε και από εκεί και πέρα είναι απόφαση του καθενός αν θα χρησιμοποιήσει αυτές τις δυνατότητες ή όχι. Αλλά πολλοί επιστήμονες λένε ότι ο άνθρωπος έχει συμπόνια, πρέπει να έχει μεγαλύτερη συμπόνια. Όλοι έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να πετύχουμε την εσωτερική ειρήνη. Και μέσω της εσωτερικής ειρήνης μπορεί να επιτευχθεί η πραγματική ειρήνη στον κόσμο. Μόνο μέσα από την εσωτερική ειρήνη. Γιατί η οργή και ο φόβος είναι συναισθήματα που είναι αδύνατον να οδηγήσουν στην ειρήνη. Έχω λοιπόν δεσμευτεί για τρία πράγματα. Πρώτον, την πρόθεση της ενότητας των 7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Πάντοτε τα λέω αυτά. Στο θεμελιωδώς είμαστε όλοι οι ίδιοι. Στο, σε, δεύτερο, στο, δεύτερο επίπεδο υπάρχουν διαφορές εθνικότητας, χωρών, θρησκευτικές διαφορές, χρώμα, χρώματος, αλλά και μέσα σε μια ίδια ομάδα υπάρχουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι, οι μορφωμένοι και οι αμόρφωτοι, πολλές, πολλές διαφορές. Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα οφείλονται ότι δίνουμε υπερβολική σημασία στις δευτερεύουσες ε, διαφορές μεταξύ των οποίων είναι οι θρησκευτικέ συγκρούσεις, οι εθνικές συγκρούσεις. Αυτού του είδους τα προβλήματα δεν λύνονται δια της βίας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μόνο αν προχωρήσουμε στο βαθύτερο επίπεδο όπου όλοι είμαστε άνθρωποι και τότε καταλαβαίνουμε ότι το δικό του πρόβλημα είναι και δικό σου αν επιτύχει αυτός, επιτυγχάνω και εγώ. Είμαστε όλοι μαζί. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στην Ήπειρό σας, έχει ξεπεράσει πολλές συγκρούσεις, πολλές ζωές που χάθηκαν στο όνομα των εθνικών συμφερόντων. Και τώρα προχωρήσαμε στο κοινό συμφέρον. Αυτό είναι καταπληκτικό. Πάντοτε εκφράζω, μιλάω για το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάποια στιγμή θα πρέπει να διαδοθεί στην Αφρική, η Αφρικανική Ένωση κατά κάποιο τρόπο. Μερικοί ονομάζουν, το ονομάζουν Παναφρικανισμό. Αυτό Πιστεύω ότι αν αυτό επεκταθεί στην Αφρική θα περιοριστούν πολλά προβλήματα, αλλά και στην Ασία. Πραγματικά λοιπόν αισθάνομαι ευγνώμων, αισθάνομαι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ για να απευθυνθώ, για να μιλήσω στο κατά πρόσωπο με πρόσωπο στα μέλη του Κοινοβουλίου. Έχω εδώ φίλους από πολύ παλιά. Ένας Γερμανός που είναι πολύ παλιός μου φίλος. Ένας πραγματικά μεγάλος υποστηρικτής της υπόθεσης του Θιβέτ, που είναι μια δίκαιη υπόθεση. Πολιτικά δεν επιδιώκουμε την απόσχηση. Η πρώτη μου δέσμευση λοιπόν είναι η προώθηση της έννοιας ότι και τα 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι ίδιοι. δεύτερη είμαι θρησκευτικός, είμαι θρήσκος, είμαι βουδιστής. Για να είμαι πιο ακριβής, είμαι μαθητής, οπαδός των μεγάλων δασκάλων. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι είμαι φιλόσοφος στοχαστής. Για μένα οι μεγάλοι αυτοί δάσκαλοι στην ουσία είναι επιστήμονες. Κάποιες, κάποιες γραφές έχουν απορριφθεί. Η διδασκαλία του βουδισμού λένε ότι αντιβαίνει τη λογική. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να τα απορρίψουμε μερικά πράγματα. Οι μοναχοί, οι οπαδοί δεν πρέπει να δέχονται τη διδασκαλία μου δια της βίας, αλλά μετά από σκέψη και έρευνα. Ως λοιπόν βουδιστής καλόγερος, μοναχός, ευθύνη μας είναι να προωθήσουμε την αρμονία όλα τα θεσμικά όργανα, όλοι οι θεσμοί μεταφέρουν το ίδιο μήνυμα. Τη συμπόνια, τη συγχώρεση, την ανοχή. Όλοι, τα, όλοι οι θρησκευτικοί θεσμοί αυτό προωθούν. Υπάρχει λοιπόν κοινό έδαφος, κοινή πρακτική και σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να οικοδομήσουμε πραγματική αρμονία με αμοιβαίο σεβασμό μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον. Η Ινδία είναι ένα ζωντανό παράδειγμα. Όλες οι θρησκευτικές παραδόσεις συνυπάρχουν. Κατά καιρού υπάρχουν προβλήματα, αλλά εν γέννη επικρατεί μια εξαιρετική αρμονία. Η Ινδία είναι μια δημοκρατική χώρα και υπάρχει αρμονία. στον υπόλοιπο κόσμο, σε άλλες περιοχές υπάρχουν πολλά προβλήματα. Είναι λοιπόν πολύ εφικτό να μπορεί κανείς να συνυπάρξει με αρμονία αυτή. Η τρίτη μου δέσμευση αφορά το Θιβέτ. Είμαι από το Θιβέτ. Από την πολιτική έχω ήδη αποσυρθεί. Είμαι λοιπόν δεσμευμένος στην διατήρηση του πολιτισμού του Θιβέτ που τη συνήθως την περιγράφω ως πολιτισμό της ειρήνης, της μη βίας. Δεύτερον, τις γραφές του Θιβέτ. διαπιστώνω ότι η γλώσσα, η γραφή του Θιβέτ είναι καλύτερη για την περιγραφή της λογικής δεν είναι ούτε τα η Ινδική γλώσσα, ούτε τα Κινέζικα, ούτε τα Σανσκριτικά. Αυτό αξίζει να διατηρηθεί, αυτή η γλώσσα και η γραφή. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διατηρήσουμε τις γνώσεις μας. Οι αρχαίοι δάσκαλοι δίδαξαν μόνο στα θηβετικά την βουδιστική παράδοση και κατόπιν το περιβάλλον. Ένας οικολόγος από την Κίνα έγραψε ένα άρθρο που ανέφερε τις επιπτώσεις που προσ... τι προσφέρει το υψίπεδο του Θιβέτ σε σχέση με την υπερθέρμανση του παλί, πλανήτη. Μίλησε για το Βόρειο Πόλο, τον Νότιο Πόλο και είπε ότι το Θιβέτ είναι ο τρίτος πόλος. Από εκεί καλύπτεται σχεδόν ολόκληρη η Ασία. Έτσι λοιπόν η προστασία του περιβάλλοντος του Θιβέτ δεν αφορά μόνο τα εκατομμύρια των Θιβετιανών αλλά τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων. Αυτές οι τρεις λοιπόν δεσμεύσεις μου, είμαι 81 ετών, ίσως τα επόμενα 15 χρόνια ή 20 χρόνια θα έρθει η στιγμή να αποχαιρετήσω, να αποσυρθώ. So. Οπότε, αυτά είχα να σας πω και τώρα θα ακούσω τις ερωτήσεις σας και θα αρχίσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Μπρόκ, σας ευχαριστώ πολύ. Δέκα και πέντε θα είναι η, ε, το όριο για την αναχώρηση. Όμως όλα αυτά τι σημαίνουν. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που ζήτησαν να παρέμβουν. Έχουμε πολλούς. Ε, ο κύριος Τένο και πάνω. Παρακαλώ να περιοριστείτε σε ένα λεπτό όλοι σας. Θέλω να μπορέσουν το δυνατόν περισσότεροι αγορητές να παρέμβουν θα ήταν σωστό και δίκαιο να το κάνουμε αυτό. Και από τους συντονιστές ζητώ να παρέμβουν για ένα λεπτό, να τηρήσουν αυτό το όριο, ώστε να μπορούν οι περισσότεροι να παρέμβουν. Ο κύριος Πρέδε έχει τον λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να καλωσορίσω την αγιότητά σας. Είναι μεγάλη τιμή για μας η παρουσία σας εδώ. Είναι πολύ επίκαιρη η επίσκεψή σας γιατί αυτή την εβδομάδα συζητήσαμε στην Ολομέλεια την θέση της Κίνας στην διεθνή σκηνή. Νομίζω ότι παρά τις προσπάθειες τις οποίες έχει κάνει η οικονομική κυβέρνηση για την οικονομική ανάπτυξη, η Κίνα είναι μια μεγάλη δύναμη και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να σεβαστεί τα δικαιώματα των πολιτών και να προχωρήσει στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και τον σεβασμό των μειονοτήτων. Γι' αυτό και υποστηρίζουμε τους Θηβετιανούς στην αναζήτησή τους για τη διατήρηση της ταυτότητάς τους, του πολιτισμού τους, του πολιτισμού της ανοχής και της μη βίας. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Ο κύριος Κάννα. Είναι πιο δύσκολο για μένα αν συγκεντρώσετε τις ερωτήσεις. Ah, stay in my brain. Για, καλύτερα, τα θυμάμαι καλύτερα ένα-ένα. Okay, then next question. Mr. <laughs> Khan is ready. Tenok. Mr. Σας καλωσορίζω στο Στρασβούργο, λέει ο κύριος Καν. Σας καλωσορίζω και εξ ονόματος της ομάδας των σοσιαλιστών για την εξαιρετική δουλειά την οποία κάνετε, για το μήνυμα ειρήνης το οποίο εκπέμπεται και για την σωστή εκπροσώπηση του λαού του Θιβέτ. Αν μπορώ μία ερώτηση. Πολλοί από εμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχούμε ε, για τη βία που ασκείται εις βάρος της ε, μειονότητας της μουσουλμανικής των Ροχίνγκα. Η Χανσουνκή η οποία είναι γνωστή η εικόνα της ε, δημοκρατίας δεν έχει καταδικάσει τις παραβιάσεις αυτές στη Βυρμανία. Θα ήθελα λοιπόν να μας διαβεβαιώσετε ότι οι βουδιστές στη Βυρμανία που έχουν προχωρήσει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις θα τιμωρηθούν. Δώδεκα you How many questions? ερωτήσεις είναι πάρα πολλές. Oh, τρεις το I ο κύριος Φαμπάλεν παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πώς είπατε? Thank you. Thank you. Ο κύριος Τάνοκ. Αγιότατε. Πανάγιε. Σας καλωσορίζουμε εξ ονόματος της ομάδας μας ε, των Ευρωπαίων Μεταρρυθμιστών ε, και συντηρητικών. Πάντα ήμασταν φίλοι των Θηβετιανών. Πάντα ασκούσαμε επικρίσεις ε, στη δημοκρατία της Κίνας όταν προσπαθούσαν να καταπιέσουν τον πολιτισμό του Θηβέτα. Ε, στο αναφέρεται το δικαίωμα για την αυτονομία και την αυτοδιάθεση του. Όμως ε, Καλωσορίζω τα δικά σας λόγια ότι η ακαιρεότητα της Κίνας δεν διακυβεύεται με κατακαιρματισμό. Είσαστε ένας άνθρωπος της ειρήνης με όραμα. Σας σεβόμαστε ως θρησκευτικό ηγέτη. Έχετε ένα το αίσθημα του χιούμορ και όσο μεγαλύτερος, όσο γυρεότερος γίνεστε, τόσο και πιο αστείος γίνεστε στα όσα μας εκθέτετε. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μακρύ ταξίδι της ζωής σας. Μακάρι να μπορέσετε να ζήσετε πολλά χρόνια για την παγκόσμια ενότητα, την ειρήνη και την αρμονία που σας εύχομαι να δείτε να υλοποιούνται. Thank you. Μπορούμε να πάρουμε άλλη μια ερώτηση τώρα. Εσείς κύριε Φαμπάρεν, ευχαριστώ. Φυσικά συμφωνώ απόλυτα με τα όσα ανέφερε ο κύριος ε, Τάνοκα. Έχω μια ερώτηση, ε, Πανάγιε ερώτηση. Όλη τη ζωή σας προσπαθούσατε να βρείτε τρόπους συζητώντας και διαπραγματευόμενος με τους ε, Κινέζους για να λυθούν ειρηνικά οι διαφορές όχι ζητώντας ανεξαρτησία αλλά πολιτική ελευθερία και αυτονομία υπάρχει κάποιο άνοιγμα επίσημα από πλευρά των Κινέζων προς αυτήν την κατεύθυνση είναι απόλυτα κλειστή νομίζω σε σχέση με αυτή την ερώτηση θα μπορούσαμε να ε, πάρουμε άλλη μία ακόμα αν υπάρχει μία παρόμοια άλλη μία επιτρέψτε μου να απαντήσω basically... Ουσιαστικά πιστεύω ότι η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας έχοντας το ίδιο κομμουνιστικό κόμμα με το ίδιο σύνταγμα στην πραγματικότητα υπάρχουν κάποιες αλλαγές ε, κατά, σε σχέση με τα τελευταία 40 χρόνια δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό υπάρχουν κάποιες αλλαγές και μετά έπειτα σήμερα οι βουδιστές, οι βουδιστικοί πληθυσμοί στην Κίνα περίπου 400 εκατομμύρια. Υπάρχουν πολλοί Κινέζοι βουδιστές που αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η παράδοση και η θρησκεία του Θιβέτ είναι αυθεντικά στοιχεία, αξιόλογα και θέλουν να μάθουν από αυτή την παράδοση. Και μετά έχουμε και τους ανώτατους ηγέτες της Κίνας. Μεταξύ αυτών υπάρχουν ενδείξεις ότι συνειδητοποιούν και αυτοί ότι η πολιτική τους ε, όπως είχε ακολουθηθεί δεν, ήταν, δεν είναι ρεαλιστική. Υπάρχει κάποια αλλαγή λοιπόν σε σχέση με την οτροπία και τη σκέψη τους πώς να επιληθούν πολλά άλλα προβλήματα, ακόμα και το ζήτημα του Θιβέτ. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις γι' αυτό. Ωστόσο όμως στην καθεστική ατάξη στο κατεστημένο είναι απόλυτα κατανοητό ότι εξακολουθούν να τηρούν τη σκληρή γραμμή την οποία εκφράζουν και εκθέτουν. Βασικά λοιπόν υπάρχει ελπίδα ουσιαστικά. Υπάρχουν ενδείξεις ελπίδας και είναι σημαντικό ο έξω κόσμος, ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το δει αυτό. Δηλαδή, σε σχέση με την προσπάθεια να υπάρξει βοήθεια για το μέλλον, για το μέλλον και της Κίνας. Δηλαδή, με, με επικοδομητική κριτική που καμιά φορά είναι αναγκαία να εκφράζεται, αυτή τη στιγμή ακόμα και οι σκληροπυρηνικοί Κινέζοι αντιμετωπίζουν κάποια διλήμματα. Πώς να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα και να τα επιλύσουν. Σε μια τέτοια συγκυρία, σε μια τέτοια χρονική στιγμή, η κοινή γνώμη, παγκόσμια κοινή γνώμη και η στάση της μπορεί να επηρεάσει αυτούς τους ανθρώπους κάπως. Αντίθετα με τη δεκαετία του 60 ή 70 που αδιαφορούσαν για το τι πίστευε ο έξω κόσμος ε, και ποια ήταν η άποψη των πολιτών εκτός Κίνας. Αυτή είναι η απάντηση προς την πρώτη ερώτηση και στην τρίτη και τέταρτη ερώτηση. Τώρα, σε σχέση με το ότι όταν πρώτα άκουσα για μουσουλμάνους σε σχέση με την Βυρμανία και την, τις διώξεις αυτών των μουσουλμάνων ήμουνα στη Βόσιγκτον, με ρώτησαν σχετικά και εξέφρασα και είπα ότι θέλω να συμμεριστώ ή θέλω να πω σε αυτούς τους ε, πληθυσμούς, των βουδιστικούς πληθυσμούς, αν έχετε προβλήματα με κάποιους μουσουλμάνους, φυσικά να, θα έπρεπε να σκεφτείτε, να αναλογιστείτε το πρόσωπο του Μπούντα. Τι θα έκανε. Αν βρισκόταν εκεί ο Βούδας, σίγουρα θα λάμβανε υπόψη και θα προστάτευε τους αδερφούς ε, και τις αδερφές μουσουλμάνους και μουσουλμάνες στη Βυρμανία. Και αρκετά, ε, είχα την ευκαιρία να το πω αυτό και κατά κάποιο τρόπο μια και είναι πάρα πολύ περίπλοκο αυτό το θέμα, νομίζω ότι για αρκετά μεγάλη περίοδο υπήρξε, ας το πω έτσι, σιγή για αυτό το θέμα. Δεν υπήρχαν τοποθετήσεις γι' αυτό. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να τοποθετείται κανείς ανοιχτά και να μιλάει γι' αυτό και να τοποθετείτε κατά αυτών των φαινομένων και των διώξεων. Μετά, σε σχέση με τους μουσουλμάνους, από την 11η Σεπτεμβρίου που συνέβη αυτό το τρομοκρατικό πλήγμα, προβαίνω σε επαφές με διάφορους μουσουλμάνους, έχω επαφές και γνωρίζω ότι οι μουσουλμανικές κοινότητες που στη Λάσα είναι πάρα πολύ ήρεμη και ειρηνική και πολύ ευγενική και ποτέ δεν δημιούργησε οποιοδήποτε πρόβλημα. Έχω και πολλούς φίλους στο Λαντάκ της Ινδίας και έχω πολλούς φίλους που είναι μουσουλμάνοι και είναι πάρα πολύ ακέραιοι και σωστοί άνθρωποι. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε σχέση με κάποιους που λένε ότι υφίσταται τρομοκρατία βουδιστική και υπάρχουν βουδιστές τρομοκράτες ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι μεμονωμένοι εκπροσωπούν όλους τους βουδιστές και δεν είναι λοιπόν ε, τρομοκράτες οι υπόλοιποι βουδιστές αν κάποιος ε, ε, άσκησε βιοπραγίες κατά των μουσουλμάνων δεν είναι οι βουδιστές στο σύνολό τους τρομοκράτες έναντι των μουσουλμάνων. Και τώρα κατά τους τελευταίους μήνες πιο πρόσφατα με πολλές, σε πολλές αφορμές ε, στη ΣΥΠΑ αλλά και στην Ευρώπη λέω και αναφέρω ότι υπάρχουν βουδιστές ε, τρομοκράτες αναφέρεται και μουσουλμάνοι τρομοκράτες είναι πάρα πολύ αρνητικό αυτό. Οποιοςδήποτε θέλει να ενταχθεί σε μια βία παράταξη και να, κάνει, να ασκήσει βία, δεν μπορεί κανείς αυτό να το επεκτείνει στους υπόλοιπους και να λέει ότι είναι οι άλλοι που φταίνε όλοι για τους βουδιστές ή για τους ε, μουσουλμάνους. Οι ίδιοι οι οποίοι είναι τόσο βίαιοι δεν είναι αυθεντικοί εκπρόσωποι των ε, θρησκειών τους, του, της μοαμεθανικής θρησκείας ή του βουδισμού. Τζιχάντ σημαίνει να ξεκινήσει κανείς να ελέγχει τις δικές του, ε, ε, τα δικά του αισθήματα και τις δικές του, τα δικά του συναισθήματα, ώστε να μπορεί να έχει την αυτοκυριαρχία και να είναι τελειότερος. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι είναι τζιχαντιστές λένε είναι μουσουλμάνοι, δεν είναι μουσουλμάνοι χρησιμοποιούν την επίκληση της θρησκείας αλλά δεν είναι θρησκευόμενοι και δεν ασκούν τη δική τους θρησκεία όπως θα έπρεπε. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε λοιπόν μεταξύ αυτών των πραγμάτων. Δεν θα πρέπει να γενικεύουμε και να λέμε ορίστε όλοι οι μουσουλμάνοι είναι τρομοκράτες ή όλοι οι βουδιστές είναι ε, επικίνδυνοι. Καθόλου και πραγματικά πιστεύω γι' αυτό για τους βουδιστές τρομοκράτες όταν υπάρχουν κάποια τέτοια δημοσιεύματα στο περιοδικό Time στην Αμερική και με φωτογραφίες και αναφέρεται ορίστε βουδιστές τρομοκράτες αισθάνομαι μεγάλη αμηχανία και αισθάνομαι πραγματικά ότι με πιέζει, καταπιέζει αυτό δεν είναι σωστό βουδιστές τρομοκράτες Μεγάλη αμηχανία αισθάνομαι γιατί αυτό είναι ψεύδος, δεν αληθεύει, δεν υπάρχουν βουδιστές τρομοκράτες. Και από την άλλη πλευρά, όταν έχουμε και όποτε έχουμε την ευκαιρία να συναντόμαστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εκφράζουμε αυτό και να το λέμε ο ένας τον άλλον. Υπάρχει διαφορετική δυνατότητα προσέγγισης. Να συνέρχεται κανείς με λόγιους, με ιεροσπουδαστές, να βλέπει ποιες είναι οι τα κοινά σημεία και ποιες είναι οι διαφορές. Υπάρχουν διαφορές, ε, υπάρχουν διαφορές ε, ενιολογικά και στην προσέγγιση. Κάποιοι λένε είναι δημιουργός ο Θεός του κόσμου. Εμείς δεν έχουμε την έννοια ως βουδιστές του πλάστη του κόσμου, του δημιουργού του κόσμου. Και πρέπει να ε, δούμε λοιπόν σε σχέση με αυτό ότι κάποιοι λένε ότι είμαστε αμαρτωλοί μια και δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και δεν το δεχόμαστε αυτό. <clears throat> Θα πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με έναν μεγάλο φίλο τον οποίο έχω και τον οποίο συναντώ όποτε συναντώμαστε ε, μου έλεγε ότι ορίστε εγώ ε, θεωρώ ότι εσείς ο εκπρόσωπος ο ανώτερος θρησκευτικό εκπρόσωπος και μετά από ημέρες συζητήσεων μια φορά ανέφερε και είπε ότι είμαι ε, είναι έτοιμος να μπορέσει να πάει στον παράδεισο πλέον και η δική μου αναφορά ήταν ότι μπορεί κανείς να πάει σε διάφορα σημεία και όχι υποχρεωτικά στον παράδεισο Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, λόγω του ότι υπάρχουν ενοιολογικές διαφορές ε, δεν παίζουν ρόλο αυτές, ε. δεν είναι αυτές οι σημαντικές, τα σημαντικότερα στοιχεία. Ο στόχος είναι να υπάρξει η αναγνώριση και ο σεβασμός των αξιών και των αρχών για την αξία, για παράδειγμα, της συμπόνιας. Λέγεται όλοι δημιουργηθήκαμε από, έναν, από τον Θεό, έναν Θεό Όλοι λοιπόν είμαστε πλάσματα αυτού του Θεού. Ακόμα και εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Λοιπόν, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί το δυναμικό της αγάπης και της κατανόησης. Η φιλανθρωπία, η συμπόνια, οι θρησκείες με όλες τις, ε, ε, σε όλες τους τις τάσεις ε, αυτό λένε. Και η συνάντηση και η άσκηση των πραγματικών αυτών αρχών Σύμφωνα με τη δική μου πείρα, η συνάντησή μου για παράδειγμα με τον επίσκοπο τούτου και σε αυτές τις συζητήσεις που είχα μαζί του και τον Τόμας Μάρτον δεν γνωρίζω το όνομα ενός καθολικού μοναχού στη Βαρκελόνη ο οποίος όμως μοναχός πέντε ολόκληρα χρόνια έζησε ως ε, μοναχός ε, στο κελί του με πολύ λίγη τροφή ε, ως ερημίτης με ελάχιστη τροφή. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω και τον ρώτησα ποια ήταν η πρακτική στη ζωή σου. Ήταν η πρακτική της αγάπης είπα, είπε στην απάντησή του και βλέπουμε ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα αυτό που ανέφερε. Η αγάπη, η πρακτική, η άσκηση της αγάπης. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από τον καθολικισμό υπάρχει μια τέτοια μαρτυρία και με άλλους μουσουλμάνους που είναι εξαιρετικά άτομα. Συναντώντας λοιπόν τέτοιους ανθρώπους που ουσιαστικά ασκούν αυτές τις αρχές ανταλλάσσοντας ε, τις ε, δικές τους ε, βαθύτερες εμπειρίες και βιώματα. Κάνει πολύ σημαντικό το να κατανοήσει κανείς τον άλλον. Και αυτό είναι η τρίτη δυνατότητα των προσκυνημάτων προσκυνήματα σε Άγιους τόπους και η δυνατότητα διαλογισμού και αναστοχασμού μαζί με αυτούς. Και αυτό είναι πάλι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ο διαλογισμός για να μπορέσει κανείς να ανυψωθεί ψυχικά. Και με την αρχαία παμπάλε, παμπάλες ρίζες της α, ε, α, ε, χριστιανικής συριακής ε, εκκλησίας και θρησκείας. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο διαλογισμός και η βαθιά, ε, ο βαθύς στοχασμός, θρησκευτικός στοχασμός και στην Ινδία σε σχέση με την άσκηση αυτών των αρχών και για τους βουδιστές ε, ε, μερικές ομάδες χριστιανών που υπάρχουν εκεί, χριστιανοί αλλά και Ινδουιστές ε, που προσχώρησαν και τοπικοί εκπρόσωποι του τοπικού πληθυσμού και επί 20 ε, λεπτά υπήρχε ενσυγή διαλογισμός. Ήταν κάτι πολύ ε, επικοδομητικό και θετικό ε, για να υπάρξουν τα πνευματικά θετικά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Όποιοι λοιπόν, όποιοι άνθρωποι έχουν τέτοιες πεπιθήσεις, ας προσπαθήσουν να δημιουργήσουν όλο και περισσότερες συναντήσεις ε, και επαφές, ανταλλαγές σε όλα τα επίπεδα με τους υπόλοιπους είναι σημαντικό εκδηλώσεις τέτοιες στη Γαλλία, στις Βρυξέλλες, ε, σαν αυτές που έγιναν. Και μετά στη Συρία επίσης, στο Ιράκ, ε, στη Λιβύη και στο Πακιστάν και Αφγανιστάν σε κάποιο βαθμό επίσης. Και οι Σουνίτες και οι Σιήτες ε, μουσουλμάνοι προς την ίδια κατεύθυνση πώς είναι δυνατόν να σκοτώνουν, να δέχονται να δολοφονούνται άνθρωποι. Ασύλλητο, αδιανόητο αυτό. Γιατί η ζωή και η ε, αξία της πρέπει να προστατεύεται. Και πρέπει να ασκείται η αγάπη. Δεν είναι δυνατόν να μπορεί να δεχτεί κανείς ότι θα μπορεί να σκοτώνονται άνθρωποι, να δολοφονούνται άνθρωποι. Είναι αδιανόητο κάτι τέτοιο. Όσοι άνθρωποι έχουν θρησκευτικές πεπιθήσεις, ακόμα και εκείνοι που δεν έχουν θρησκευτικές πεπιθήσεις και οι αθεϊστές ακόμα, θα πρέπει να αγωνίζονται για να διασώσουν και να προστατεύσουν τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ευχαριστώ. Αυτά είχα να σας πω. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. 30 δευτερόλεπτα, πέντε άνθρωποι που θέλουν να πάρουν το λόγο και μετά η αγιότητά του θα κάνει τις καταληκτικές του παρατηρήσεις. Κατάλογο κατάλογος των ονομάτων, των ομιλητών. Σας ευχαριστώ αγιότατε που προσήλθατε. Θερμό καλωσορίσατε και από την ομάδα μας, την Ελεύθερη Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Έχω τις εξής παρατηρήσεις. Ε, αισθάνομαι αμήχανος και με... Α, δεν μπορώ να σας δω. Είναι πολύ μικρό το μικρόφωνο και γι' αυτό... Γι' αυτό έσκυψα, ναι πραγματικά με πλήττουν, με συγκλονίζουν οι αυτοπυρπολήσεις των Θηβετιανών ε, και που βρίσκονται στην ε, προσπάθεια να διατηρηθεί, να διαφυλαχθεί η παράδοση και η ταυτότητα του Θηβέτ. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αυτό το γεγονός των αυτοπυρπολίσεων. Δεύτερη ερώτηση. Ανησυχώ για την εξόριξη ουρανίου στο Θηβέτ που έχει τεράστιες οικολογικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εδώ θα ήμουν ευγνώμων για ένα σχόλιο που θα μπορούσατε να μας κάνετε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μας που είσαστε εδώ. Εκπροσωπείτε το σύνολο του λαού του Θιβέτ. Με βλέπετε εδώ στο βάθος. Εσείς εκπροσωπείτε λοιπόν τον Θιβετιανό λαό και Αυτά τα 60 χρόνια μη βίαιης αντίστασης έχετε δώσει το παράδειγμα. Εσείς δεν θέλετε να φύγετε από την Κίνα, θέλετε όμως να ενωθείτε με την ανθρωπότητα. Μία ερώτηση. Τι δεν κάνουμε σαν Ευρωπαίοι και δεν βοηθάμε έτσι την υπόθεση του Θιβέτ. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε ελπίζοντας ότι θα δημιουργήσουμε κάποια στιγμή και σε αυτό το κοινοβούλιο ένα intergroup για το Θιβέτ. Η τελευταία ερώτηση είναι πράγματι μία αντίσουμε εμεί σαν βουλευτές. Ο κύριος Μποργέζιο. Ευχαριστώ την αγιότητά σας για την παρουσία της εδώ. Συναντηθήκαμε στους διαδρόμους την ώρα που ε, φτάνατε εδώ, σας καλωσόρισα και αμέσως μιλήσατε για το δικαίωμα των λαών στην ελευθερία. Σας ευχαριστώ για αυτά τα λόγια. Είναι ένα μάθημα που δίδεται στην κρατούσα πολιτική τάξη στην Ευρώπη, ιδιαίτερα τους μεγάλους ηγέτες της τάξης της πολιτικής που ε, ντρέπονται να συναντήσουν μια τόσο υψηλή θρησκευτική προσωπικότητα. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι κάθε επιτυχία και πάντα θάρρος. Παναγιώτατε, κάποιοι ευρωβουλευτές είχαν την ευκαιρία στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση 200, για το Θιβέτ 250 από πολλές χώρες. Ερώτηση. Το ψήφισμα που υποστηρίζαμε έλεγε πάντα να μεριμνήσουμε ο διάλογος μεταξύ της Κίνας και των Θιβετιανών και των εκπροσώπων των Θιβετιανών να μπορεί να διεξαφεί. Βλέπετε μια δυνατότητα να μπορεί να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος. Εγώ δεν είμαι θρήσκα, παρόλα αυτά όμως έχω πάντα να κερδίσω όταν μπορώ να συζητήσω μαζί σας. Θα ήθελα να σας μεταφέρω κάτι το οποίο πιστεύω. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι αυτό το οποίο είπατε ε, την πραγματικά ηθική εξουσία, την εξουσία δηλαδή της ηθικής καλύτερα κανένας δεν μπορεί να την αγοράσει. Ότι έκαναν ερωτήσεις όλοι οι συνάδελφοι. Εγώ απλώς θέλω να σας πω ότι στηρίζω ολόθερμα τα 7 σημεία σας για το Θιβέτ. Ελπίζω ότι θα υπάρξει ένας πραγματικά θαραλέος ε, πολιτικός ηγέτης της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας, ο οποίος θα καθίσει δίπλα σας και θα συζητήσετε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Now, very, very sad. When... Για τους αυτοπυρπολούμενους είναι κάτι πάρα πολύ θλιβερό. Εκφράζω τη θλίψη μου για αυτό το τρομερό θλιβερό γεγονός. Ταυτόχρονα όμως από την άλλη πλευρά είναι τόσο δραματική αυτή η μορφή πράξης που πρέπει να την μας υποχρεώσει να μας κάνει να πάρουμε σοβαρά και αυτήν και τα πράγματα τα οποία επικαλούνται οι αυτοπυρπολούμενοι. Ουσιαστικά η θέση μου είναι πάρα πολύ δύσκολη, διληματική. Δεν μπορώ να υποστηρίξω τις αυτοπυρπολήσεις. Αν ήμουν δημόσια εναντίον, πολλοί, πολλά μέλη οικοί και συγγενείς αυτών των ατόμων θα θεωρούσαν, θα αισθανόντουσαν μεγάλη θλίψη. Ούτως ή άλλως θα ήταν, ήταν τόσο συντετριμένοι και με τη δική μου καταδίκη ακόμα περισσότερο θα θλιβόντουσαν. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η που όπως ήδη προανέφερα έχουμε και το περιβάλλον στο Θιβέτ. Επειδή βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο και σε πολύ ξηρό ε, ε, υποξηρασία όσον αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες, είναι πάρα πολύ ευάλωτο, εύθρωτο, σε υψηλό υψόμετρο και με ξηρότητα, ξηρό, ε, ξηρή ατμόσφαιρα, αν υπάρξει κάποια ε, βλάβη οικολογική, περιβαλλοντική, θα απαιτηθεί πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να επουλωθεί. Και μετά επίσης ε, το θέμα της προστασίας του υψηπέδου και οικολογικά που δεν αφορά 6 εκατομμύρια άτομα ως κατοίκους της περιοχής αλλά δισεκατομμύρια άτομα παγκόσμια. Και ένας από τους πρώην πρωθυπουργούς ε, κατά τη διάρκεια της θητείας του πολλές από τις πλημμύρες που είχαν σημειωθεί στην ίδια την Κίνα είχε αναφέρει και είχε πει ότι θα έπρεπε να υπάρξει μικρότερη αποψήλωση των δασών για να μην σημειώνονται αυτές οι πλημμύρες, αυτά τα φαινόμενα. Υπήρχαν όμως φαινόμενα διαφθοράς τότε και ποιο ήταν το επόμενο. Η κινέζικη κυβέρνηση και οι τοποθετήσεις της φαίνεται ότι υπάρχει κάποια εντύπωση, κάποια τάση να υπάρξουν διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις. Όμως, απλά θέλουν να επικοινωνήσουν με μένα ως άτομο. Άτομο μεμονωμένο, τον Δαλάη Λάμα, όχι ως εκπρόσωπο των Θηβετιανών. Και ποτέ δεν χρησιμοποιείται ο όρος Θηβετιανή κυβέρνηση οι Κινέζοι όταν ε, μας κατηγορούν χρησιμοποιούν ε, τέτοια ορολογία. Εμείς όχι. Ταυτόχρονα όμως εμείς ποτέ δεν χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους ε, όρους. Μας κατηγορούν οι Κινέζοι και λένε εσείς χρησιμοποιείτε τον όρο το μεγαλύτερο Θιβέτ. Τι είναι εκείνο το οποίο αναφέρουν και λένε. Πρώτον, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχουν πάνω από 100.000, 150, 160.000 πρόσφυγες ε, ε, που πρέπει να μεριμνήσουμε για αυτούς, να υπάρξει μέριμνα για αυτούς και για τη στέγασή τους, ε, την κατάρτισή τους, εκπαίδευσή τους και για την προαγωγή των θηβετιανών πολιτιστικών αξιών και της θηβετιανής παράδοσης. Πρόσφατα μπορεί κανείς να πει ότι αυτά θεωρούνται ανεδαφικά. Το 2011 αποσύρθηκα 100% όχι μόνο εγώ αλλά και από 400, 400 χρόνια, 400 αιώνες παράδοσης που 4 ε, αιώνες παράδοσης που ε, τέλειωσαν και τώρα μελλοντικά στο μέλλον θα έχουμε την δημοκρατία ως σύστημα που θα ακολουθούμε. Δημοκρατία, ένα καλό σύστημα. Και έτσι λοιπόν και η δική μας ε, κοινότητα θα πρέπει με βάση τις αρχές της δημοκρατίας ε, να κυβερνάτε. Τώρα, σε σχέση με την κυβέρνηση της Κίνας, ε, λαμβάνουν πολύ περισσότερο υπόψη αυτά τα οποία έχω εγώ αναφέρει από ότι εγώ ο ίδιος. Και σε σχέση με Κινέζο φίλο, αν θέλετε πραγματικά να εκφράσετε κάποιο ενδιαφέρον ή να εκφράσετε για την μετεμψύχωση του Δαλάη Λάμα ε, το ενδιαφέρον σας θα έπρεπε το Κομμουνιστικό Κόμμα να αναγνωρίσει την ε, ιδιότητα της μετεσάρκωσης και δεύτερον σε σχέση με την Κίνα να αναγνωριστεί ότι υπάρχουν κάποιοι υψηλοί ε, λάμας. Οι ίδιοι λοιπόν οι Κινέζοι δέχονται τις ε, αρχές ε, του Βουδισμού και ακολουθούν ακόμα και τις αρχές του Θηβετιανού Βουδισμού. Και σε σχέση με αυτά, όποιος πιστεύει στην αναγέννηση, οι Κινέζοι κομμουνιστές θα έπρεπε να προσπαθήσουν να βρουν ποια είναι η μετεμψύχωση του Προέδρου Μάο. Και τότε θα μπορούσαν να πούν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια μετεμψύχωση του Δαλάη Λάμα. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει λογική σε αυτά τα επιχειρήματα. Στο μέλλον λοιπόν ο Δαλάη Λάμα δεν θα έχει και δεν θα μπορεί να έχει πολιτική εξουσία. Oh, I want, Θέλω να κάνω έκκληση. Πάντοτε λέω όταν συναντώ ε, κάποια κοινοβουλευτική ομάδα, οπουδήποτε, ζητώ κυρίως να συζητηθεί το πρόβλημα της οικολογίας. Και τότε λέω, επισκεφθείτε το Θιβέτ. Βρείτε Κινέζους οικολόγους και από κοινού επισκεφθείτε τις σε αυτές περιοχές και συντάξτε μια έκθεση. Ίσως και η κυβέρνηση της Κίνας να χρειάζεται κάτι τέτοιο, μια ρεαλιστική, πραγματιστική έκθεση ε, εμπειρογνωμόνων, μια ανεξάρτητη έκθεση. Ίσως αυτό βοηθήσει. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, όταν ε, εκφράζετε την ανησυχία σας για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την θρησκευτική ελευθερία. Ίσως οι Κινέζοι να αντιδράσουν διαφορετικά. Οπότε έχετε την ευκαιρία να πείτε ας ταξιδέψουμε προς τα εκεί για να δούμε εμείς οι ίδιοι την κατάσταση. Επισκέψεις από το εξωτερικό και ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα βοηθήσουν πάρα πολύ πιστεύω, τουλάχιστον στο μυαλό του λαού του Θιβέτ. Θα τους ενθαρρύνει. Αυτό είναι το αίτημά μου. Και κατόπιν η ομάδα υποστήριξης του Θιβέτ είναι απαραίτητη. Είναι πολύ σημαντική. αυτή η σκληρή γραμμή, των, οι Κινέζοι που έχουν τη σκληρή γραμμή δεν θα συζητήσουν το θέμα του Θιβέτ παρά μόνο εάν δεν διαπιστώσουν ότι το θέμα του Θιβέτ δεν θα φύγει από το τραπέζι. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Thank ευχαριστούμε πολύ. Αρχιότατε. Αδερφές και αδερφοί που αντιμετωπίζουν τόσα δεινά και Φυσικά θα πρέπει να εκφράζει κανείς την ανησυχία του γι' αυτό και είναι καμιά φορά σημαντικό να εκφράζει κανείς αυτά τα συναισθήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Παναγιώτατε που προσήλθατε εδώ και βρήκατε το χρόνο να μπορέσετε μεταξύ των πολύ σημαντικών θεμάτων που σας απασχολούν να έρθετε και να ασχοληθείτε και μαζί μας ε, και για τα επίπεδα των, της διαφοροποίησης ε, που παραμένουν όλοι οι άνθρωποι όμως ε, ανθρώπινα όντα είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που θα πρέπει να θυμόμαστε αυτό που μας δώσατε. Είναι σημαντικό αυτό για να κατανοήσουμε καλύτερα την πολιτική ζωή και να πάμε σε μεγαλύτερο βάθος. Υπήρξε μεγάλη πίεση που ασκήθηκε για να ακυρωθεί αυτή η συνεδρίαση σήμερα το πρωί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικαίωμα να συναντά όποιον επιθυμεί και δεν μπορεί κανείς αυτό να της το αφαιρέσει. Και γνωρίζω, γνωρίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε και με την Κίνα που είναι σημαντικότατη χώρα και για την πολιτική της One China Policy. Πρέπει όμως να μπορούμε να μιλάμε και για τις αξίες ε, και τις αρχές αυτές με θρησκευτικού ηγέτες και κανείς δεν μπορεί να το αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα από εμά. Και αυτό ανήκει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που είχατε και προσήλθατε σε εμά. Σας ευχαριστώ, το εκτιμώ ιδιαίτερα. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη στεναρή στάση σας. Ευθύς εξ αρχής την εκτιμώ. Διότι εσείς υιοθετήσατε στεναρότατη στάση με βάση ηθικές αρχές ε, σε σχέση με αυτή τη συνεδρίαση. Εμείς ακολουθούμε αυστηρότατα τις αρχές της μη βίας. Απόλυτα με μη βίαιο τρόπο από συμπόνια δίνουμε ε, την προσπάθεια αυτής της, ε, αυτού του αγώνα και θα πρέπει έτσι να μπορέσει να στεφθεί, με, να, να επιτύχει. Και στο Θιβέτ ε, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα της αυτοπυρπόλησης και ο αγώνας, η μάχη μας με αυτόν τον τρόπο λέγεται δεν θα ε, παράξει αποτελέσματα. Το κάνουν αυτό λόγω του ότι βρίσκονται σε απόγνωση. Εσείς όμως με τη στάση σας, με την ηθική σας θέση και στάση είναι πιο σημαντική αυτή από ότι χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ.